Okay, colleagues, we have a long list of votes to do, so we are going to make a start. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ήθελα να καλωσορίσω κάποιους εκπαιδευόμενους ε, μεταφραστές οι οποίοι βρίσκονται στο πίσω μέρος της αίθουσας σας καλωσορίζω, ξέρω πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που καλείστε να κάνετε και εγώ είχα εκπαιδευτεί ε, για αυτό το επάγγελμα. Ελπίζω να παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι μετά από τις ψηφοφορίες έχουμε άλλα δύο θέματα με προσκεκλημένους ομιλητές Το ένα είναι η ανάληψη ευθύνης για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και το δεύτερο χρηματοδότηση της αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών για το τι θα γίνει μετά το COP21. Γι' αυτό θα ήθελα οι συνάδελφοι να είναι παρόντες ανάμεσα στις 4 και 4 και στις 6.30. Σχετικά με τις κανονικές ψηφοφορίες είπαμε ότι το 16 η έκθεση δηλαδή για τη συνάντηση κορυφή στην ανθρωπιστική θα είναι το τελευταίο προς ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε με το 17 Κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμα την, τον κατάλογο ψηφοφοριών. Are people happy? They haven't got their voting list through. Is that the problem? Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. You vote against uh, your Maybe there could be one copy at least for the coordinator of the EPP, then the others could follow. Ίσως να δώσετε ένα αντίγραφο στον συντονιστή του ΕΛΚ και οι άλλοι να τον ακολουθούν. Okay, well, we have one copy for the EPP. Now we can do it. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τεστ τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Η ηλεκτρονική δοκιμαστική, το αναλαμβάνω. Ψήφισαν 18 από τις 21 κάρτες. Εγώ δεν ψήφισα. 20 τώρα. Καλώς δουλεύει το σύστημα. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Το ΕΛΚΑ έχει τον κατάλογο τώρα. Θα ξεκινήσουμε με το 17. Η έκθεση Μπεσέρα για την κατάσταση στη Μεσόγειο σε σχέση με τα θέματα της μετανάστευσης. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Κοιτάξτε, τα έχω μπλέξει λιγάκι. Βλέπω τον κατάλογο εδώ, αλλά δεν είναι ο σωστός κατάλογος. Λοιπόν, δεκτή τροπολογία 2. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3, ποιοι είναι υπέρ. Α, όχι βέβαια, έχει καταπέσει η τροπολογία 3. 12. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 12. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13. Προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα μάλλον καταπίπτει. Το δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος του δεύτερου τμήματος της 16 ψηφίζεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 18. Ποιοι είναι υπέ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απερίφθη ή μάλλον ή δεκτή ή απερίφθη θα δούμε, αλλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά για να δούμε ακριβώ τι έχει συμβεί. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη με μικρή διαφορά. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ, συγγνώμη, 23 υπέρ, 23 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, 24 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 24. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 31. Υπέρ. Κατά Αποχές. Απερίφθη νομίζω. Α, έτσι κι αλλιώς έχει καταπέσει, δεν πειράζει. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 37 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 38 υπέρ κατά αποχές απερίφη... 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές απερίφη... 41 Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 41. The, vote is closed. Απερίφθη. Α, ο κύριος Πρέντα το αποφάσισε. Λοιπόν, 42 υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 46 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 47 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 α όχι 48 άρχεται η ψηφοφορία α για 48 ψηφίσαμε α απερίφθη 49 τώρα υπέρ κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 49. Τέλος. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Α, ε, τι, δεκτή, 51, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 55, υπέρ, κατά, αποχές, Πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 55. Ελέγχουμε, ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 6. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 59 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 60 υπέρ, κατά, Αποχές δεκτή. Απερίφθη μάλλον, απερίφθη. 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ 75 υπέρ, κατά, αποχές. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 75. Τέλος της ψηφοφορίας δεκτή. Have some confusion here. Amendment 77. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 78. Δεκτή με μικρή διαφορά 81 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 81 τέλος δεκτή 84 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη νομίζω, αλλά θα υπάρξει έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 87. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 87. Τέλος της ψηφοφορίας. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή, νομίζω. Όχι, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 88. Πέρας της ψηφοφορίας δεκτή. Γι' αυτό οι συντονιστές καλύτερα να σηκώνουν ψηλά τα χέρια τους παρακαλώ. Το 89 υπέρ. Κατά. Αποχές Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος και εδώ για την 89. Πέρας της ψηφοφορίας ε, απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 91 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 92 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 93 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το 93 τέλος απερίφθη 94 υπέρ κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 94. Πέραση της ψηφοφορίας. Δεκτή. Λοιπόν, τελική ψήφος. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. 21 υπέρ, 1 κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ την κυρία Μπεατρίς Μπεσέρα Μπαστερετσέα. Πάμε τώρα στο 18. Κοινοί κανόνες για την εξωτερική διάσταση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Εδώ θα είναι σύντομη η ψηφοφορία. Δύο τροπολογίες, η έκθεση Χόιμπουχ, ένα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, δύο υπέρ, σε δύο τμήματα μάλλον. Το πρώτο τμήμα, ναι, λοιπόν ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, δεκτή, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρω, έλεγχος για το δεύτερο τμήμα, τέλος, δεκτή. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος. Δεκτή. 21-1-1. Περνάμε τώρα σε μια μεγαλύτερη ψηφοφορία για το 19. Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και στην Ένωση. Ο κύριος Φρουτζούλητσα είναι ο εισηγητής. Υπάρχουν αρκετές συμβιβαστικές τροπολογίες. Ξεκινάμε με την παρήθμ 1. Ποιοι είναι υπέρ της 1. Α, η Λόλα έχει ζητήσει το λόγο. θα ήθελα να μην παραλείψουμε την ψηφοφορία των προφορικών τροπολογιών. We need two members in this committee. Does another member object? Λοιπόν, ε, διαφωνεί κάποιος. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ε, διαφωνεί μάλλον κάποιος, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει η ψηφοφορία αυτή. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά απερίφη. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απερίφη. Έξι υπέρ. Α, κάτι ξέχασα. Πω πω ξέχασα. Πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική 4. Πρώτα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 7. Δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στην 34 πηγαίνουμε τώρα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 34. Τέλος. Δεκτή. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 44 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 44 πέρας της ψηφοφορίας δεκτή 45 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 45 υπέρ. Πέρα της ψηφοφορίας δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Ξανά από την αρχή λέει η 47 με ενοχλεί ο κύριος Πρέντα. 47 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έλεγχος ηλεκτρονικά για την 47. Απερίφθη έτσι κι αλλιώς. 48. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 49. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Πενήντα έξι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εξήντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 60. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο της νομοδότησης. Ψηφίσατε όλοι. Λοιπόν, διορθώθηκε το τεχνικό, ψηφίζουμε, τέλος, δεκτή, 22 υπέρ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φραντζούλητσα. Okay, we move to item 20 now, which is the firstly the oral question. σημείο της ημέρα της διάταξης για την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις κρίσης. Εδώ έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, μιας και πρόκειται απλώς για προφορικό ερώτημα χωρίς τροπολογίες. Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή. Ψήφισαν όλοι. Ένας λείπει. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα. Πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία όμως, θα ήθελα να ανακοινώσω δύο διορθώσεις που έγιναν χτες το βράδυ στον κατάλογο ψηφοφοριών. Στη δεύτερη σελίδα, ε, τροπολογία 59, αυτή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι καταπίπτει αν εγκριθεί η συμβαστική F. Δεύτερη διορθώση, η τροπολογία 10 εμφανίζεται δύο φορέ. Φυσικά θα ψηφίσουμε μόνο μία φορά. Και αυτό το λάθο βρίσκεται στη σελίδα 5. Και παρόλο που σα το είπαμε, σίγουρο ότι κάποιο θα μου το υπενθυμίσει ότι θα φτάσουμε, αλλά εν περιπτώσει για να μην υπάρξει σύγχυση. Όταν φτάσουμε λοιπόν για πρώτη φορά στη τροπολογία 10 πριν την 1, θα ψηφίσουμε. Ωραία, τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτά, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία γιατί στο προφορικό ερώτημα, ξεκινώντα από τη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Μάλλον εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. 52 συγγνώμη. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά.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 κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83, την πραγματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα, για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, για το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 83, ένα ψηφοφορίας. της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 84. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88. Έχει αποσυρθεί. Και πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποσχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποσχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποσχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποσχές εγκρίνεται συμβιβαστική B, Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20... Τροπολογία 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 34 τμηματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα τελική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίστε Everybody Αν ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορίας και με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλους τους κοιόδης για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν. we now move to... Περνάμε τώρα στο σημείο 21. Εφαρμογή των συστάσεων του 2010 για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη. Η συγγήτρια Λεόλα και εδώ έχουμε κάποιους ε, συμβασμούς, συμβαστικές τροπολογίες και περνάμε στην συμβαστική α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική β, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τη συμβαστική β, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 13. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 22. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 14 ψήφοι υπέρ 9 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στην εισηγήτρια. Okay. So um, just to say, Amendment 49, we're voting now. Τροπολογία. Τώρα 49. Ψηφίζουμε την τροπολογία του κυρίου Γκερέρο Σαλόμ για την παγκόσμια διάσκεψη για τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Έχει γίνει μία αλλαγή. Αποσύρθηκε η τροπολογία 49 από τον κύριο Βέντα. Ψηφίζουμε τώρα το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. amendment 43. In Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν. Μάλλον όχι. Αποσύρθηκε. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Κατά. Αποχές. Δεν μου δείχνατε τι θέλετε. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 88. Αρχίζουμε. Α, μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Πέρας. Ναι, δεν καταλαβαίνω το πώς σηκώνετε τα χέρια σας, τι θέλετε. Λοιπόν, 92, δύο τμήματα. 90, με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 90 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μάλιστα. Και εδώ είναι σαφές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 109. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 117 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Συμβιβαστική 117 μάλλον. Πέρας. Όταν αργείτε να σηκώσετε το χέρι, με μπερδεύετε. Δεύτερο τμήμα της 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128. Καταπίπτει. Ψηφίζουμε τώρα τις συντηλικές σκέψεις. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία 6. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι σοσιαλιστέ. Ψηφίσατε υπέρ. Εγκρίνεται τότε. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 26. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35. 36. Μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται των παραθέσεων. Ψηφίζουμε τώρα τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών. Στην παράγραφο 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην υπο... γνωμοδότηση της Υποεπιτροπής ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Είχαμε και μερικές εποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή. Και νομίζω πως τώρα τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε, ήρθαν οι εμπειρογνώμονες. Okay, colleagues, we're going to make a start. We gave our, our guest a little bit time to arrive because we, we finished Κάναμε ένα μικρό διαλυματάκι για να δώσουμε το χρόνο στου ε, προσκεκλημένου μα να έρθουν γιατί αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε. Ελπίζω τώρα οι εκπαιδευόμενοι διερμηνοί μα να βρουν πιο ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω από του εκπαιδευόμενου διερμηνεί, μάλιστα να του βοηθήσουμε να ακούσουν τη διερμηνία. Έχουν ακουστικά, Επομένω μπορούν να μελετούν του διάφορου γλωσσικού συνδυασμού, τις διάφορες γλώσσες προς τις έχουμε διερμηνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βρουν και τα λάθη μα. Να περάσουμε στο 21 τη μέρης της λοιπόν. Οι συντονιστε είχαν ζητήσει να γίνει μια συζήτηση επί της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της πρόοδου που έχουν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη της όσον αφορά τη λογοδοσία ε, στην χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας για το 2015. Αυτή η ε, έκθεση έχει εκδοθεί πριν από την Σύνοδο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία. Τα ζητήματα αυτά της λογοδοσίας και της χρηματοδότησης τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας. Όπω πολλέ φορέ έχουμε συζητήσει και άλλα θέματα οικονομική πολιτική των κρατών μελών. Γι' αυτό χαίρομαι που έχουμε μαζί μα εμπειρογνώμονε με ε, μεγάλη και ε, εμπειρία που μπορούν να μας μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα. Έχουμε τέσσερις ομιλητές. Κυρία Μαρινίσεν από την ε, Γενική Διευθύνση ΤΕΦΚΟ, Φαντερπόλ από την Οργάνωση Κονκόρτ, ε, ένας εκπρόσωπος της 11.11.11 μιας φλαμανδικής οργάνωσης ε, για την ανάπτυξη και τον υπεύθυνο για θέματα ε, δικαιοσύνης και ανάπτυξης και τον κύριο Έντουμπερκ από τον ΟΑΣΕ ο οποίος παλαιότερα εργαζόταν και στην Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Νορβηγίας. Έχει επίση επαγγελματική εμπειρία στην Παγκοσμία Τράπεζα. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Μαρινίσεν, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι είναι πολύ ε, χρήσιμο να ξεκινήσουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτήν την έκθεση για τη λογοδοσία. Θα ήθελα και εγώ όπως πρότεινε η Λίντα να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν. Όπως γνωρίζετε, η έκθεση για το 2015 καλύπτει δύο άξονες. Πρώτα απ' όλα εξετάζει ε, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι οικονομικές αναφορές, οι αναφορές για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας από το 2002 και μετά. Και επίσης εξετάζει την ετήσια έκθεση του 2014 που κάλυπτε τα τελευταία 14 χρόνια και η οποία μας επέτρεψε να προετοιμαστούμε για την συνάντηση στην Αντίσα Μπέμπα τον Ιούλιο. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε ε, επί τη βάση των απαντήσεων σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που στέλναμε στα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη τα τελευταία 13 χρόνια, βασιζόταν στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας αρχικά και με την παρόδο του χρόνου καλυφθήκαν και άλλα ζητήματα όπως η εμπορική συνεργασία, η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, η χρήση των ε, πόρων των εθνικών, η έρευνα και άλλα. Επομένως τα ερωτηματολόγια θα έλεγα ότι ε, έγιναν πολύ πιο πλήρη και προσπαθήσαμε επίσης να εξετάσουμε και κατά πόσον είμαστε αποτελεσματικοί θέτοντα στόχου και κοιτώντα αν του πετύχαμε. Από του 41 στόχου που είχαμε θέσει, 23 από αυτούς επιτεύχθησαν, είτε βρίσκονται σε καλό δρόμο και 9, για 9 από αυτούς τους στόχους ε, έχουμε μια μερική επιτυχία. για άλλους στόχους, κυρίως εκείνους που αναφέρονταν σε ποσοτικούς στόχους αναπτυξιακούς της χιλιετίας, δεν τα έχουμε καταφέρει. Αυτό μας δίνει μια γενική εικόνα του που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ε, εντοπίζει σε ποιες περιοχές τα καταφέρνει καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αποτελεσματική και σε ποιος όχι και τόσο το θεωρούμε ένα χρήσιμο εργαλείο για τη λογοδοσία. Το χρησιμοποιούμε τα τελευταία 13 χρόνια. Βεβαίω, ένα αντίστοιχο σύστημα δεν είχε ε, υιοθετηθεί στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών μέχρι τη σύνοδο της Αντισάβετα. Τώρα ξεκινάμε σε παγκόσμιο επίπεδο να δημιουργείται ένα τέτοιο σύστημα λογοδοσία, Δεν γνωρίζουμε ακριβώ ε, θα διαμορφωθεί, αλλά είναι κάτι στο οποίο έχουμε συμφωνήσει. Στο οποίο έχει συμφωνήσει η κοινότητα. Στην έκθεση του 2015 διαπιστώνουμε ότι οι τομεί στους οποίους είμαστε ιδιαίτερω επιτυχεί ήταν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και η ενίσχυση του χρήση των εθνικών πόρων, και αύξηση των επενδύσεων. Οι άμεσε ξένε επενδύσει επίση έχουν αυξηθεί τα τελευταία 13 χρόνια στι ε, χώρε μέσου εισοδήματο, αλλά στι ε, λιγότερο αναπτυγμένε ε, κατώτερου μέσου εισοδήματο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι ε, επίσης ε, σίγουρα σα ενδιαφέρει το ζήτημα των νέων τρόπων χρηματοδότησης, ιδιαίτερα των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και πολλέ φορέ. Στον τομέα των παραδοσιακών δωρεών τη άμεση αναπτυξιακή βοήθεια. Και παρά το γεγονό ότι τα τελευταία χρόνια το λέμε διαρκώ ότι η άμεση αναπτυξιακή βοήθεια μειώνεται, συνεχίζει να έχει τον πρώτο ρόλο, την καθεδρία. Είναι γνωστό ότι ο στόχος του 0,7% δεν επετεύχθη, αλλά η δέσμευση να τον πετύχουμε επαναβεβαιώθηκε στην Αντεσάβεβα. Όσον αφορά την βοήθεια την εμπορική. Εδώ ε, έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Το ίδιο ισχύει και για την βοήθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το 2013 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν ως ε, ενισχύσεις για τον τομέα του εμπορίου. Παραμένει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ανοιχτή αγορά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η... Έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εμβασμάτων και ψάχνουμε να δούμε πώς αυτά θα μπορούσε να μειωθεί. Και ενθαρρύνουμε επίσης, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων αναπτυσσόμενων χωρών στα ερευνητικά μας προγράμματα. Και συχνά προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με τις αναπτυσσόμενες χώρες για να βελτιωθεί η διαφάνεια, ιδίως στα προγράμματα που από κοινού διοργανώνονται ε, με αυτές τις χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τι πρέπει, να τι πρέπει να γίνει στο μέλλον, πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε κατά πόσον, να φροντίζουμε μάλλον να πετύχουμε τους ε, ποσοτικούς, τους οικονομικούς στόχους ε, και τους σχετικούς με τους SFDG και τους σχετικούς με την αναπτυξιακή βοήθεια. Όπως έλεγα, δημιουργείται σιγά σιγά ένα σύστημα λογοδοσίας στο επίπεδο του ΟΗΕ και θα πρέπει να φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο με τον οποίο εξέταζε ετησίως ε, την οικονομική επίδοση της αναπτύξης της βοήθεια, βοήθειας. Να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη γνώση και να την περάσουμε στο παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε τελικά το σύστημα που θα φτιαχτεί στον ΟΗΕ να είναι το καλύτερο δυνατό. και μετά να προσαρμόσουμε και εμείς το δικό μας σύστημα ε, εκθέσεων και λογοδοσίας ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές που θα έχουμε αντιοποιήσει. Να υπάρχει ένα ε, μοναδικό σύστημα για τη λογοδοσία και την αξιολόγηση του κατά πόσο πετυχαίνουμε και τους στόχους για το θεματολόγιο 2030 και τους SDG. Επομένως οποιαδήποτε ε, σχόλιο ή παρατήρηση ή πρόταση έχετε να κάνετε για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το σύστημα λογοδοσίας στο μέλλον είναι ευπρόσδεκτη. Μπορείτε να μας στείλετε και γραπτό τις προτάσεις σας. Ή φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και διαζώσεις. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ υλικό και πολύ τεκμηρίωση εδώ. Ο επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Βαντερπούλ, από την Φλαμανδική μη κυβερνητική 11 ο οποίος θα μας μιλήσει για την πλατφόρμα των ΜΚΟ που λέγεται Concord. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο στην Επιτροπή σας σήμερα πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ομιλώ εκ μέρους της Concord λοιπόν που είναι η πλατφόρμα αν θέλετε μέσα από την οποία εκπροσωπούνται εκατοντάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπεύθησαν και στην Άντισα Μπέμπα στην τρίτη διάσκεψη και θα ήθελα να πω ότι από πλευράς όλων αυτών των οργανώσεων που ήσαν εκεί ότι αισθάνθηκαν μια κάποια απογοήτευση ακόμα και το ακρόνιμο FFD σημαίνει ουσιαστικά Failure to Finance Development το FFD και αυτή την αίσθηση την ένιωσαν όσοι ήσαν εκεί παρόντες και δικαιολογημένα. Βλέποντας το τι προήλθε Στην ουσία υπάρχουν πάρα πολλά λόγια υποστήριξης αν θέλετε της διαδικασίας αλλά παρόλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αντίστοιχο με τις φιλοδοξίες που έχουμε για το πλαίσιο το αναπτυξιακό και τη χρηματοδότησή του που συμφωνήθηκε στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο και για τους νέους στόχους αηφορίας που θα πρέπει να ισχύσουν από το 2013 και μετά και δεν είναι αντίστοιχο των προσδοκιών έτσι και αλλιώς των πολιτικών μας. Δεν υπάρχει απαιτούμενη επαρκής χρηματοδότηση από πλευράς των εθνικών προϋπολογισμών σε επάρκεια Δεν υπάρχει διεθνής, αν θέλετε, επίπεδο αναγνώρισης των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, δεν υπάρχουν κοινέ μέθοδοι αξιολόγησης ε, και των διαδικασιών αλλά και του παρόντος εμπορικού συστήματος που ακολουθείτε. Δεν έχουν ε, ε, υπάρξει αναλύσεις σε βάθος και φοβάμαι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Νομίζω όμως ότι υπήρξε και το φόρουμ συνέχειας των συζητήσεων, κάτι το οποίο ήταν θετικό. Οι συζητήσεις όπως είπα θα συνεχιστούν. Είναι κάτι το θετικό αυτό. Αυτό το φόρουμ λοιπόν υψηλού επίπεδου το οποίο συμφωνήθηκε μετά το τέλος της πρώτης διάσκεψης κρατάει τη συζήτηση ζωντανή. Αυτά ήθελα να πω πάρα πολύ σύντομα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα περάσουν σε επίπεδα λεπτομέρειας υψηλότερα. Αλλά για τις ελεγόμενες εκθέσεις ε, υπευθυνοποίησης, αν θέλετε, νομίζω ότι η πρώτη έκθεση που κυκλοφόρησε ήταν αρκετά πληροφοριακή η έκθεση σημειώνει ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος σε σχέση με την κινητοποίηση εθνικών εσωτερικών πόρων με στόχο την βελτίωση των, και την στήριξη των φορολογικών μηχανισμών κτλ. Αλλά δυστυχώς δεν λέγει το τι θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Ε, σχετικά με τα θέματα της διαφάνειας των μεγάλων επιχειρήσεων, των ομίλων επιχειρήσεων μετά από το LuxLeaks. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση με το Country by Country Reporting, ε, έκθεση ανά χώρα ε, και στην οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων σαν παράδειγμα δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία να προβλέπεται να γίνουν. Η έκθεση λοιπόν πάρα πολύ σύντομα τώρα ενισχύει ε, κάποιους από τους κανόνες οι οποίοι ίσχυσαν. Ταυτόχρονα όμως η Ευρώπη μπλοκάρει κάποιες συζητήσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Εθνών και τους μηχανισμούς εφαρμογής των αποφάσεων αυτών σε σχέση με τους στόχους τώρα η κυρία Μαρέντσεν από την Επιτροπή το είπε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Δανία, στις σκανδιναβικές χώρες δηλαδή, όπου για μια μακρά περίοδο θεωρείται ότι ήταν πρωτοπόροι σε σχέση με την προσπάθεια επίτευξης των στόχων, οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει γιατί είναι κάτι που υπονομεύει την αξιοπιστία της Ένωσης μιας και θα συνεχίσουμε σε σημαντικό επίπεδο διαπραγματεύσεων για το κλίμα σύντομα και η Ευρώπη αμφισβητεί την ίδια της την αξιοπρέπεια εδώ. Έχουμε προβλήματα και σε άλλους τομείς στον, στο εμπόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το έκθεση κατανομής ευθυνών λοιπόν η έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται σε επιμέρους διμερείς συμφωνίες εταιρικές συμφωνίες γεν, γενικότερα γενικευμένα μάλλον προγράμματα προτιμήσεων εμπορικών όλα αυτά είναι μέσα τα οποία εν μέρη μόνο χρησιμοποιούνται για να τονώσουν, για να λειτουργήσουν σαν μοχλός για την επίτευξη των στόχων, για την ανάπτυξη. Ε, αυτά τα οποία απαιτεί ε, από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, βλέπουμε ότι έχουν υπάρξουν εξαιρέσεις από τις εμπορικές προτιμήσεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέσο πλέον αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι η βοήθεια για το εμπόριο, το Aid for Trade. Εδώ οι εξελίξεις θα πρέπει να επανεξεταστούν γιατί υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις τις οποίες θέτουν ερευνητές και για τη χρηματοδότηση του κλίματος εισαγωγικά. Οι αριθμοί είναι σαφείς από το 12 μέχρι το 13,56 δις αλλά υπάρχουν πολύ υψηλότερε προκλήσεις, δεν υπάρχει μεθοδολογία αναφορά των ενεργειών αυτών και δεν υπάρχει διεθνώς συμπεφωνημένη μεθοδολογία για την βοήθεια για την αντιμετώπιση ή τη μετρίαση των συνεπειών. Υπάρχει μια ανισότητα από ό,τι νομίζουμε εμεί στήριξη ανάμεσα στην προσαρμογή από τη μία και την μετρίαση των συνεπειών από την άλλη. 43% μετρίαση και το υπόλοιπο για την αντιμετώπιση και εξέλιξη. Νομίζω ότι απαιτείται υψηλότερο ποσοστό για τις προσαρμογές. Τελευταίο σημαντικό θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τώρα στη διάθεσή της περισσότερα μέσα στην παρούσα φάση για την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων προσαρμογής και μετρίασης των συνεπειών και μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με την επιχειρηματική ευθύνη, την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Υπάρχει το θέμα το οποίο άπτεται και ε, των μη χρηματοδοτικών μέτρων και των υπολείπων ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για να υπάρξει σωστή ε, και κατανοητή λειτουργία καταμέτρησης ή υπολογισμού αν θέλετε των μέτρων αυτών θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα επιπλέον και να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε τα πράγματα όταν διαπιστώνονται κάποιες τέτοιου είδους αρνητικές πλευρές. Δεν έχω άλλες παρατηρήσεις. Έτσι βλέπουμε εμείς σαν Κονκόρντ την έκθεση αυτή ευθύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρναμε τώρα στον Τόρβα Μαρία Ράιντινγκ που ειδικεύεται σε ζητήματα φορολογικού δικαίου. Μας έχετε φέρει και κάποιον πίνακα, βέβαια δεν μπορούμε να δούμε τα χρώματα για την ασπρόμαυρη εκτύπωση. Α, όχι, μόλις μου έφεραν και την έγχρωμη εκτύπωση. Πολύ ωραία. Θα μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε σε θέματα φορολογικού δικαίου και φορολογικής δικαιοσύνης. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη, μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά ήρθα εδώ για να σας μιλήσω για φορολογικά ζητήματα, αλλά και για ιδιωτική χρηματοδότηση και για το χρέος. Καταρχάς ε, για τα φορολογικά ζητήματα. Θα ήθελα να πω ότι όσοι από εσάς ήσασταν στην ε, Αντισαμπέμπα στην ε, διάσκεψη θα θυμάστε ίσως ότι κύριο κομμάτι της συζήτηση ήταν εάν οι αναπτυσσόμενε χώρες έχουν το δικαίωμα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όταν τα παγκόσμια φορολογικά πρότυπα διαπραγματεύονται εκεί. Επίσης θα ξέρετε ίσως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε έντονα για το θέμα αυτό πολλές φορές και σε μια έκθεσή του από την Έλλη Σλάιν που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τον Ιούλιο με μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία. Ποιο είναι το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ένα σύστημα όπου όσα και κάποιες φορές ε, οι G20 διαπραγματεύονται και αποφασίζουν τους κανόνες και τα πρότυπα για την παγκόσμια φορολόγηση για όλους μας. Αυτό σημαίνει ότι 140 αναπτυσσόμενες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την διαδικασία. Τη διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται αποφάσεις για παγκόσμιους κανόνες. Έχουμε δηλαδή από τη μία τους ε, υπεύθυνου της πολιτικής αυτής, τον ΩΣΑ και την G20 και τους υπόλοιπους που απλά πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες που έχουν αποφασιστεί σε συναντήσει τι οποίες δεν ήταν προσκεκλημένοι. Ίσως είναι δύσκολο να καταλάβουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη που σε γενικές γραμμές θεωρούν ε, αυτούς δημοκρατικές χώρες υπερασπίζονται ένα τέτοιο σύστημα το οποίο αποκλεί άλλες χώρες από τη λήψη αποφάσεων σε φορολογικά ζητήματα. Τα φορολογικά ζητήματα είναι κεντρικό σημείο μιας δημοκρατικής χώρας είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ενεργότατο ρόλο στην Αντισαμπέμπα έτσι ώστε να διατηρηθεί το status quo. Και υπήρξε η πρόταση δημιουργίας ενός παγκόσμιου φορολογικού ε, σώματος υπό την αιγύδα των Ηνωμένων Εθνών, κάτι το οποίο απερίφθη. Μάλιστα διάβασα την έκθεση για τη λογοδοσία και εξεπλάγει, διότι στη σελίδα 31 Ευρωπαϊκή Επιτροπή γράφει ότι είναι μια πολύ σημαντική δέσμευση που θα ενισχύσει την συμμετοχή των αυτοσόμενων κρατών στην αφορολογική συνεργασία. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπλόκαρε τη συμμετοχή αυτών των χωρών. Και το επιχείρημα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε και στους G7 και στους G20 και στον ΩΣΑ. Και αυτά είναι τα φόρα από τα οποία αποκλείονται οι αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι προφανές πιστεύω πως χρειάζεται να αλλάξει στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Ε, τώρα, σχετικά με το χρέος, να σας πω ότι είδαμε κάποιες πολύ θετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών όπου έχουν αναπτυχθεί κάποιες αρχές σχετικά με τον υπεύθυνο δανεισμό. Και δημιουργήθηκε και μια διαδικασία για μηχανισμό έλεγχου του χρέους, του διεθνούς χρέους. Χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρέους θα έχουν κάπου να καταφύγουν, κάτι το οποίο δεν ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτός ο μηχανισμός θα χρησιμεύσει ε, στο να αντιμετωπίσει αυτά τα επικίνδυνα ταμεία, τα, τα ταμεία όρνια όπως λέγονται, vulture funds. Βέβαια, παρότι αυτές οι πρωτοβουλίες βρήκαν την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο με το τελευταίο του ψήφισμα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, αλλά και ε, στο παρελθόν ε, υποστηρίχθηκαν και από τα κρατη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και από τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ως ε, φορέας αρνήθηκε να συμμετάσχει στις συζητήσεις και κάποια μάλιστα καταψήφισαν στα Ηνωμένα Έθνη την πρόταση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν σα είπα πως εξεπλάγει όταν είδα τη σελίδα 34 της έκθεσης όπου αναγράφεται ότι, ότι η δέσμευση 8 έχει τηρηθεί και η δέσμευση 9 σχετικά με τις ε, διεθνείς ε, συνεργασίες επίσης αλλά και η δέσμευση 11 για την καταπολέμηση αυτών των ε, επικίνδυνων ταμείων, των τοκοβληφικών ταμείων. Οι πρωτοβουλίες βέβαια στα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζονται, οπότε πιστεύω πως δεν είναι αργά για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συμπεριληφθεί σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Χρειάζεται διάλογος με τις αναπτυσσόμενες χώρες και αν θυμάστε στην Αντίσα Μπέμπα έγινε λόγος για διεθνή πρότυπα για τις ε, συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα βέβαια οι προτάσεις καταψηφίστηκαν και από τα αναπτυσσόμενα κράτη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλήφθηκαν δεσμεύσεις για να γίνουν διάφανες και ανοιχτές συζητήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις, ε, τα έγγραφα και τις πληροφορίες για τις συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Και ο διάλογος αυτός, εκτός από ανοιχτός, να γίνει σε διεθνές φόρουμ. Αυτό που μας εξέπληξε είναι ότι από τα 56 κράτη που δεσμεύτηκαν, λίγα από αυτά είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θετικό βέβαια είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν τώρα πιο ενεργά. Βέβαια αυτό θα ήθελαμε να το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση για τη λογοδοσία φαίνεται πως ασχολείται με αυτό το θέμα και το προσεγγίζει ως κάτι εύκολο. Όμως το blending αυτό όπως ονομάζεται είναι κάτι το πολύπλοκο και πολύ αντιφατικό. Το Παγκόσμιο Πλαίσιο για την Ανάπτυξη μετά το 2015 ζητά την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ε, την, ε, τον αντίκτυπο του blending. Και έχουν εκφραστεί μάλιστα αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά του. Ακόμα και το ελεκτικό συνέδριο έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για το blending και εξετάζοντας κάποια έργα και την προστιθέμενη αξία αυτών δεν ε, βρέθηκε αυτή η προστιθέμενη αξία και μάλιστα αμφισβητήθηκε και η αποτελεσματικότητά του και η προστιθέμενη αξία του. Και δυστυχώς λόγω λήψεων στην διοίκηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε το blending, τα ωφέλη που έπρεπε να έχει. Τώρα, αν διαβάσετε τη συνέχεια της έκθεσης, δεν θα βρείτε κάποια κριτικά σχόλια γι' αυτό. Και στη σελίδα 195 θα δείτε ότι αναφέρεται πάλι η ίδια έκθεση με λιγότερο θετικό ε, βλέμμα, όμως δεν έχει αρνητική χρειά σε γραμμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και τις συστάσεις στην έκθεση. Και τέλος, πόσο αποτελεσματική είναι η βοήθεια. Το blending επιφέρει και διάφορους κινδύνους ε, ως προς την αποτελεσματικότητα η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ενδεχομένως να παραμεριστεί από άλλους στόχους, για παράδειγμα την κερδοφορία των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το blending επίσης ε, μπορεί να επιδεινώσει ε, την κατάσταση όπου παρατηρούμε χρηματοδότηση να φεύγει από τα φτωχότερα κράτη, ακριβώς επειδή υπάρχουν προβλήματα στην ε, διαχείριση των κονδυλίων. Υπάρχουν και πολλά μάλιστα παραδείγματα ανακατεύθυνσης χρηματοδότησης από τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες στην μεταναστευτική κρίση και την αντιμετώπιση της στην Ευρώπη. Ε, εδώ θα αφαιρεθούν κονδύλια που προορίζονταν για τις φτωχότερες χώρες οι οποίες έχουν δεσμευτεί για τους ε, αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Υπάρχουν λοιπόν περισσότεροι στόχοι προς επίτευξη και λιγότερη διεθνής βοήθεια για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Σας ευχαριστώ για μια ανάλυση η οποία δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξία. Ο κ. Πέντερσεν, πολιτικός αναλυτής του ΩΣΑ. θα μας δώσει την προοπτική όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά του συνόλου των δωρητριών χωρών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Όπως ακούσατε υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες αυτή τη στιγμή στις διεθνείς σχέσεις για την ανάπτυξη και η συζήτηση πρέπει να γίνει γιατί είναι σημαντική. Να αναφερθώ στα θέματα της έκθεσης ευθύνης. Ποιος ε, θεωρεί ποιον υπόλογο και υπεύθυνο για ποιο πράγμα. Ε, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκαν στην ανάγκη στο μέλλον να υπάρχει μια τέτοια έκθεση ευθύνης η οποία να αποδίδει τον τρόπο με τον οποίο συγκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους στόχους ε, της ανάπτυξης και την προσφάτως υιοθετηθήσα ατζέντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε το τι μπορούμε να κάνουμε και το τι έχουμε κάνει. Είναι μια σημαντική έκθεση, περιλαμβάνει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αλλά βασίζεται πάντα στην πεποίθηση ότι μπορεί να αξιολογήσει κανείς το υπόλογο κάποιων ενεργειών μέσω συγκεκριμένων καναλιών σε επίπεδο προγραμματικό και όχι τόσο να μελετήσει το θέμα των επιπτώσεων δεν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις, δεν έχει μελετηθεί το τι συμβαίνει ε, επί τόπου, αλλά κυρίως σε επίπεδο προγραμματικό το τι λέγεται. Λοιπόν, δεν έφτασα ίσως ε, στο τέλος της έκθεσης αυτής των 195 σελίδων, αλλά ήδη στη σελίδα 14 υπάρχει μια σαφής παραδοχή από πλευρά της έκθεσης λέγεται ότι σε ό,τι έχει σχέση με τις υποχρεώσεις οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην επεξεργασία των πολιτικών, τότε τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά σε σχέση όμως με τα αποτελέσματα, της επιπτώσεις επιτόπου, τότε οι πολιτικές μας είναι εκτός πορείας. νομίζω ότι είναι μια ειλικρινής παρατήρηση, αυτοαξιολόγηση και εφόσον επαληθευτεί, το θέμα είναι το τι κάνουμε δημιουργούμε απλά νέες διαδικασίες κάθε φορά ή θέλουμε πράγματι να επηρεάσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να αλλάξουν με θετικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθει κανείς περισσότερα ε, για το τι αυτή η νέα μορφή ευθύνης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τη σχήμα θα έχει κάποιες από τις προτάσεις για τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο σχετικά με τους στόχους της αηφορίας που έχουμε υιοθετήσει στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Το βασικό πλεονέκτημα το οποίο έχουμε με τους στόχους αυτούς είναι ότι στην ουσία προσανατολίζονται στην αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα να υπάρξουν αλλαγές για τους πληθυσμούς και για, τους, για τον ίδιο τον πλανήτη. Μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχουν 17 στόχοι. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν 169 επιμέρους στόχοι. Είναι πάρα πολύ βέβαια. Όταν όμως κοιτάξει κανείς προσεκτικότερα τον αριθμό αυτό θα δει ότι δεν είναι πάνω από 100 το μόνο σε εισαγωγικά. Μόνο 100 από τους 169 αφορούν ακριβώς κάποιες επιθυμητές βελτιώσεις. Υπάρχουν τέτοιες επιθυμητές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς της ατζέντα για την αηφορία. Αν θέλω να είμαι αισιόδοξο, για πρώτη φορά έχουμε θα έλεγα ένα σαφέστατο πρόγραμμα κοινών αποτελεσμάτων για το τι αλλαγές θέλουμε να προκαλέσουμε μέσω ακριβώς αυτών των 100 στόχων με συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και σε σχέση με τον έλεγχο της υπευθυνότητας και για μας και για τους εταίρους μας. Και όχι τόσο στις διαδικασίες είτε στα νέα όργανα, στα νέα μέσα που προτάθηκαν από ορισμένου ομιλητές ή αξιολόγηση των προϋπαρχουσών διαδικασιών. Ας αλλάξουμε την οτροπία, ας δούμε τι αποτελέσματα έχουμε και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα. Πρώτον θα είμαστε σε διάλογο μεταξύ μας, με την εκλογική μας βάση, με τους εταίρους μας για συγκεκριμένες αλλαγές, για πολιτικές αλλαγές. Λόγω ακριβώς και της, του καθολικού χαρακτήρα της ατζέντα για το 2030, μπορούμε να συμπεριλάβουμε στη συζήτηση και τις χώρες τις οποίες προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Τις ίδιες βασικές αρχές έχουμε την δυνατότητα να τις συζητήσουμε σε πολιτικά επίπεδα με τους λαούς, με τους ηγέτες, με κοινό πάντα στόχο. Εφόσον το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να προκαλέσουμε και κάποιες άλλες αλλαγές. Ε, το κομμάτι της διεθνούς συνεργασίας με την οποία ασχολούμε είναι η βοήθεια. Ε, εδώ έχουμε θα έλεγα ένα πολιτικό αφήγημα τους τελευταίους ε, αιώνες το οποίο έχει σαν βασικό στόχο τη μείωση της φτώχειας. Βλέπουμε γύρω μας όμως ότι και πάρα πολλοί στόχοι όπως είπε η Μαρία έχουν αρχίσει να φαίνονται στον ορίζοντα ο τομέας του αλλαγής του κλίματος, το προσφυγικό, οι φόροι, μια ολόκληρη σειρά από θέματα εντάσσονται στο ίδιο πλέον ανομοιογενές αφήγημα. Η εκλογική μας βάση, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ και των αναπτυσσομένων χωρών έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη ρητορική, αν θέλετε, του αφηγήματος αυτού από τη μία για την αηφορία και στο τι κάνουμε, ποιες είναι οι πράξεις μας στον συγκεκριμένο τομέα από την άλλη. Νομίζω ότι οι στόχοι για το 2020-2030 για την αηφορία μας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρουμε τη συζήτηση σε ένα πολιτικό επίπεδο και να αξιολογήσουμε τους στόχους και τα αποτελέσματα καθιστώντας έτσι ικανούς τους πολιτικούς να συζητήσουν ε, με σωστό τρόπο με τους πληθυσμούς για το τι θα πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Τελευταίο σημείο να πω ότι στον ΟΣΑ δύο πράγματα κάνουμε ε, που κινούμενοι προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα workshop σύντομα, ελπίζω κάποιοι από εσά να είναι παρόντες, για τον επανέλεγχο των στόχων αυτών για την Ατζέντα 2020-2030 στα πλαίσια ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης. Και δεύτερον, όσα εργάζεται ε, στα θέματα της, του επίπεδου επίσημης ε, βοήθειας για την αηφόρο ανάπτυξη. Αυτό δεν ακούγεται και πάρα πολύ ελκυστικό ε, σαν ιδέα, δεν ξέρω και πώς μεταφράζεται σε κάθε γλώσσα. Είναι όμως μια προσπάθεια του ΟΣΑ, μια απόπειρα του ΟΣΑ που λέει ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια έχει θετικά χαρακτηριστικά, έχει αποδείξει τη χρησιμότητά της τα τελευταία χρόνια, βοηθάει τους φτωχούς στις φτωχές χώρες. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χρησιμοποιείται και για νέες εταιρικές σχέσεις και ε, για τον δημόσιο τομέα και τα δημόσια αγαθά και την διαφορετική τους χρήση κτλ. Όμως οι κυβερνήσεις και οι χώρες κάνουν πολύ περισσότερα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνολικές αλλαγές. Γι' αυτό μιλάμε για total official support, συνολική επίσημη υποστήριξη και σε επίπεδο blending, σε επίπεδο ανάμιξης δηλαδή χρηματοδοτικών μέσων και σε επίπεδο εγγυήσεων και σε επίπεδο PNPs γενικά προσπαθώντας να τονώσουμε την ατζέντα για το 2020-30. Χρειάζεται η Ευρώπη ε, για να δείξει ότι μπορούμε εμείς να διατηρήσουμε σε ισχυρό επίπεδο την επίσημη αυτή μορφή βοήθειας, κατανοώντας καλύτερα και τις υπόλοιπες αυτές μορφές επίσημης συνολικής βοήθειας για την ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ενισχύσει την πορεία επίτευξης των στόχων για την αηφορία στο νέο πλαίσιο ε, στοχεύοντας το 2030. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος Μίμητσα μας έχει ενημερώσει ότι η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει το consensus για την ανάπτυξη με βάση το νέο θεματολόγιο του 2030. Έχω ζητήσει κάποια έγχρωμα ε, φυλάδια από αυτά που σας ε, μοίρασε η Επιτροπή, γιατί έτσι μπορείτε να δείτε πολύ πιο ξεκάθαρα τους διάφορους πίνακες και διάφορα γραφήματα. γιατί βασίζεται σε ένα μοντέλο μέτρησης μεγεθών που ίσως να χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Το ερώτημα που εγώ θέτω είναι αυτό το έγγραφο το οποίο ονομάζεται έγγραφο λογοδοσίας απευθύνεται σε ποιον, δηλαδή ποιος είναι υπόλογος έναντι τίνος. Καλύτερα αυτό θα ήταν, ε, καλό θα ήταν αυτό να είναι πιο ξεκάθαρο στο μέλλον. γιατί διαφορετικά θα είχαν παρουσιαστεί τα στατιστικά στοιχεία στη μία ή στην άλλη περίπτωση και ίσως χρειάζεται σε αιτήσια βάση να εξετάζουμε τέτοιες εκθέσεις για να εξετάζουμε γιατί κάποιοι στόχοι δεν επιτεύχθησαν. Λαμβάνοντα βέβαια υπόψη αυτά που μα είπε και ο ΣΑ για την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο σύστημα με το οποίο θα παρακολουθούμε κατά πόσον έχουν επιτευχθεί η SDG, η στόχη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα δώσω το λόγο στου συζητητέ με τη σειρά που το ζήτησαν. Ε, πρώτα απ' όλα στον κύριο Σίλβα, ο οποίο ήταν συζητητή για το ζήτημα τη ε, χρηματοδότηση τη αναπτυξιακή βοήθεια, και μετά στου υπόλοιπου. Πέντρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μια και έχω τη δυνατότητα να το κάνω, θα μιλήσω πορτογαλικά. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι πράγματι αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογούμε πώς εξελίσσεται η χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια και την ανάπτυξη και θα, θα μπορούμε να βασίσουμε τη συζήτησή μας στα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται στη συζήτησή μας. Ωστόσο, με αυτά που ακούσαμε σήμερα εδώ, θα πρέπει να θεωρήσουμε το αποτέλεσμα της συνόδου στην Αντισάμπεμπα απογοητευτικό. Και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρέθηκε εκεί κατάφερε να διαπιστώσει στη διεισόμαση ότι οι χώρες δωρητρίες δεν έκαναν νέες δεσμεύσεις, δεν δεσμεύτηκαν για νέα βοήθεια, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπήρξε συμφωνία για να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των κρατών του κόσμου ε, τα ζητήματα τα φορολογικά, της καταπολέμησης των φορολογικών παραδείσων και τρίτον δεν προχώρησε το ζήτημα της αναρθιάθρωσης του δημοσίου χρέους. Και στα τρία αυτά μέτωπα δεν ε, υπήρξαν θετικές εξέλιξεις με τη Σάμπεβα. Ας δούμε όμως τα θετικά της έκθεσης αυτής. Μας δίνει στοιχεία στατιστικά, αριθμητικά. Αλλά δεν προχωράει ένα βήμα παραπάνω ώστε να αξιολογήσει και να αντλήσει κάποια συμπεράσματα από τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγμα, όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Η έκθεση αυτή μας ενημερώνει ότι αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο δεν υπήρξε τόσο μεγάλη πρόοδο όσο σε άλλου. Και ότι επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καταφέρει να επιτύχει τον στόχο που είχε θέσει για το 0,7% του ΑΕΠ. Αναρωτιέμαι, αυτή η αξιολόγηση της πραγματικότητας τη σημερινή είναι δίκαιη, είναι σωστή, δομικά τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και απλώς δεν κάναμε αρκετά ή μήπως υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα, για παράδειγμα έλλειψη πολιτικής βούλησης. Έλλειψη πολιτικής βούλησης από την πλευρά των κρατών μελών. Το στοιχείο που μας δίνει αυτή η έκθεση είναι ότι κατά μέσο όρο το 0,41% ε, αρχικά και φτάσαμε στο 5,4% ε, του ΑΕΠ ε, πήγαινε για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Με άλλη λόγια είναι, ε, έχουμε στασιμότητα. ακόμα και αν κανείς κάνει τον υπολογισμό με βάση άλλα κριτήρια, με άλλη μεθοδολογία, το μέγιστο που μπορεί να φτάσει να υπολογίσει είναι 0,44%. Επομένως, και πάλι στασιμότητα. Εξηγείται ίσως αυτό με βάση την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ή επίσης τα προβλήματα των κρατών μελών της περιφέρειας, τα οποία έχουν χτυπηθεί ε, έντονα από την οικονομική κρίση και σίγουρα δεν θα μπορούσαν εκείνα να αυξήσουν τη συνεισφορά τους. Αλλά νομίζω ότι αυτή η παρουσίαση ε, της κατάστασης κρύβει το σημαντικότερο στοιχείο που είναι ότι η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γερμανική, προσφέρει με το 1,41%. Εάν εκείνοι έδιναν περισσότερα, ο μέσος όρος της Ένωσης θα ήταν πολύ υψηλότερος και θα φτάναμε πιο κοντά στο στόχο μας. Και μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία, οικονομία την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, η οποία μάλιστα εξαιτία τη ισχύω τη θα περίμενε κανείς ότι έχει μεγαλύτερες δυνατότητες. Ε, εκείνη δεν αυξάνει την συνεισφορά τη στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Επομένω, αν κανεί έδινε και αυτά τα στοιχεία, ίσω θα ήμασταν και πιο απαιτητικοί. Θέλω να σταθώ επίση σε κάτι που είπε ο πρόσωπο του ΩΣΑ το θεματολόγιο της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη μας λέει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την εστίασή μας στην, επίσημη στην εξωτερική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και να πάμε πολύ περισσότερο σε νέα ε, χρηματοδοτικά μέσα που εμπλέκουν πολύ περισσότερο τους εθνικούς πόρους. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό. χρειάζεται αύξηση ε, μάλλον δεν αρκεί μάλλον μια αύξηση των φορολογικών εσόδων. Μπορεί τα φορολογικά έσοδα σε μια χώρα να αυξηθούν, αλλά πρέπει επίσης να μας απασχολήσει αυτά τα έσοδα που εισπράττει το κράτος, που τα αξιοποιεί, πώς τα δαπανά. Και για να κάνουμε μια τέτοιου τύπου αξιολόγηση χρειαζόμαστε άλλη, άλλη μεθοδολογία. Το ζήτημα είναι να εξετάζουμε κατά πόσον οι δαπάνε που γίνονται είτε αυτέ προέρχονται από δαπάνες του κράτου από τα φορολογικά του έσοδα είτε από ιδιωτικέ επενδύσει. εάν αυτέ οι δαπάνες εάν αυτές οι επενδύσεις τελικά γίνονται προ όφελο και προωθώντα του ε, ε, στόχου ε, ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή παρουσίαση όπως και ο Πέδρο, έτσι και εγώ πιστεύω πως είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Και θα τη διαβάσω με μεγάλη προσοχή. Θέλω όμως να σταθώ σε μερικά σημεία που μου είπατε σήμερα, με τα οποία συμφωνώ σε γενικές γραμμές. Αρχίζοντας από την πρώτη παρουσίαση, να πω ότι θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κάποιες αναφορές την κινητοποίηση των εγχώριων πόρων στην έκθεση για τη λογοδοσία. Και χαίρομαι που βλέπω πως υπάρχει αναφορά στην υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Τον Ιούλιο το Κοινοβούλιο είχε ισχυρή πλειοψηφία στην Ολομέλεια στις ψηφοφορίες για την... το μηχανισμό υποβολής εκθέσεων αναχώρα. Είναι το κυριότερο όπλο μας στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Και σίγουρα κάτι ξέρουν και στον όσα γι' αυτό. Και συμφωνώ επίσης με την σημασία των εμβασμάτων. Μάλιστα, μόλις ψηφίσαμε για την σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την μετανάστευση. Και τα εμβάσματα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης. Πρέπει να βρούμε πώς θα μειώσουμε το κόστος και με χαρά μου άκουσα πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη ήταν σίγουρα μια πολύ σημαντική στιγμή, όμως πιστεύω και νομίζω πως δεν είμαι μόνη σε αυτή την αίθουσα, ότι περιμένουμε το Μάρτιο να δούμε τι θα γίνει με τους δείκτες και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τους ε, στόχους της χιλιετίας που έχουν ήδη αποφασιστεί. Βέβαια η απόφαση είναι πολιτική και η συζήτηση είναι πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα μετρήσουμε τη διαφθορά, πώς θα μετρήσουμε την απόδοση, την χρηστή ή μη χρηστή διακυβέρνηση. Και όπως είπατε κι εσείς, πιστεύω πως πρέπει να επιμείνουμε στον ρόλο του Κοινοβουλίου, ε, όχι μόνο του Ευρωπαϊκού αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Όπως είπατε και εσείς, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό εξαρτάται και από το πόσο ικανοί είμαστε εμείς να δημιουργήσουμε καλή συνεργασία με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή. Και πιστεύω πως, θέλ, πως καλό θα ήταν να μας αφήνατε να κάνουμε περισσότερα πράγματα από όσα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει και με τη διάδραση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να έχουμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί ερωτηθήκατε πριν πώς θα το καταφέρετε και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς θα καταφέρετε να συνδυάσετε για τα δύο έτσι ώστε να έχουμε συνεκτική ε, πολιτική, έναν συνεκτικό μηχανισμό παρακολούθησης έτσι ώστε να ελέγχονται τα αποτελέσματα των προσπαθειών μα Και αν δεν κάνω λάθος, Φαντεπόλ, κύριε Φαντεπόλ από την Κορτ να πω πως συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή σας ε, για την Αντισαμπέμπα. Ε, Όντως ήταν απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Και σίγουρα δεν ανταποκρίθηκε στη φιλόδοξη ατζέντα του 2020. Όπως είπε και ο Πέδρο, το σημαντικό είναι να υπάρχει από τη μία πολιτική βούληση και από την άλλη να υπάρχουν απαρκείς πόροι. Και εντάξει, Είδαμε τι γίνεται με τους ε, πόρους, τι γίνεται όμως με τις ε, δεσμεύσεις και την πολιτική βούληση. Είδαμε, όπως είπε και ο Πέδρο, ότι πολλές φορές ε, δεν φταίει η κρίση και πιστέψτε με, Ιταλίδα είμαι, ξέρω τι σας λέω. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και αν δεν καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση των προσφύγων χωρίς ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της μετανάστευσης, χωρίς να ε, αναγνωρίσουμε ότι η ανισότητα είναι το κύριο αίτιο της ε, μετανάστευσης, εάν σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε την αναπτυξιακή βοήθεια και τα διοχετεύσουμε για να αντιμετωπίσουμε την ε, μεταναστευτική κρίση, δεν θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Ίσως το λύσουμε βραχυπρόθεσμα, αλλά όχι μακροπρόθεσμα. Πάντως, για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και την συνάδελφο που αναφέρθηκε και σε άλλα πολύ σημαντικά θέματα όπως ε, ένα πραγματικά διεθνές κυβερνητικό σώμα το οποίο θα αποφασίζει επί όρις με τις υπόλοιπες χώρες. Φυσικά πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι γίνεται με τις πρωτοβουλίες αυτές για τα φορολογικά ζητήματα. Και τέλος, είπατε ότι στην έκθεση για τη λογοδοσία έγινε κάποια πρόοδος ε, σχετικά με την τεχνική και οικονομική στήριξη των αρχών των αναπτυσσόμενων χωρών. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το 2011 λιγότερο από το 1% της ανθρωπιστικής βοήθειας είχε πάει εκεί. Να σας θυμίσω και όλα τι είπε ο Πασκάλ Σεντεμάν, ο συνάδελφός σας ε, στη Νέα Υόρκη, για την αναπτυξιακή βοήθεια. Είπε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια έχει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να την αυξήσουμε. Και εάν οι αρχές είναι σε καλύτερη θέση να διαχειριστούν τους πόρους, να τους ε, συλλέξουν, τότε θα μπορέσουμε να διοχετεύσουμε 270 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Και μπορούμε να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο την διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νταβοστήρ έχει το λόγο. Επαναλάβω αυτά τα οποία είπα ο προηγούμενος ομιλητής για το τμήμα του ODA, του στόχου που έχει σαν στόχο την φοροεισπρακτική ικανότητα, τους μηχανισμούς τους φοροεισπρακτικούς των διαφόρων χωρών. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας. Υπάρχουν πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Έχω όμως κάποια προβλήματα στην προσπάθεια αξιολόγησης αυτού του εγγράφου ε, των, ε, ε, των αποτελεσμάτων των ODA και νομίζω ότι αυτό έχει σχέση και με αυτά τα οποία προείπατε. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάποια δυνατότητα διευκρίνησης ή έστω προσθήκης κάποιων στοιχείων που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τα πράγματα. Δεύτερον, είναι σαφές ότι το χρονοδιάγραμμα 2030 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και για τις μελλοντικές αξιολογήσεις. Το θέμα είναι πώς θα λάβουμε υπόψη μας τους νέους δείκτες. Μιλήσαμε για τις ε, γενικές διευθύνσεις, μιλήσαμε για τους 169 στόχους, αλλά δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας τους δείκτες που θα τους περιλαμβάνουν. Θα εγκριθούν τον Μάρτιο ίσως και θα περάσουν από τη Γενική Συνέλευση κτλ. θα βασιστούμε στο SDG 17 ή μήπως ε, θα βασιστούμε σε όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα απαιτήσει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το πώς ε, προετοιμάζετε αυτή τη δυνατότητα. Η Χάιντι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η καλύτερη ερώτηση τέθηκε από την Πρόεδρο. Σε ποιον απευθύνεται η συγκεκριμένη αυτή η έκθεση. Νομίζω λοιπόν το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να καταστήσει υπολόγους την Επιτροπή και τα διάφορα κράτη-μέλη και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να γίνεται αυτή σε εισαγωγικά η ερωτελεστία σε αιτήσια βάση γιατί μέχρι τώρα κάτι τέτοιο προφανώς και δεν είχαμε. Μπορεί όμως να είναι και ένα, θα το χαρακτήριζε ένα κοινό μέσο αυτούς τους στόχους ε, ε, μέσα στο πλαίσιο για την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα και ο ΣΑΟ, ο οποίος είναι πάντα ένας σημαντικός ε, εταίρος για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων μέσων, και μου αρέσει η ιδέα ότι το νέο πλαίσιο 2030 θα μπορούσε ακριβώς όπως είπατε να καταστεί το νέο αφήγημα το οποίο θα ξεπεράσει απλά με μονομένα τη μείωση της φτώχειας και θα αντιμετωπίσει και τα υπόλοιπα θέματα και θα τα εντάξει στην προσπάθειά μας και ευχαριστώ τον ΩΣΑ για αυτό. Σχετικά πάντως ε, με ε, την, ε, με τον, με την αξιολόγηση της ευθύνης, περιπτώσει άκουσα κάποια σωστά ερωτηματικά. Γιατί δεν έχει υποστηρίξει την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα σώμα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών που να ασχολείται με τη φορολογική δικαιοσύνη και τα γενικότερα θέματα φορολογίας. Έχει τεθεί το ερώτημα αυτό, αλλά εγώ η ίδια δεν το έχω κάνει ακόμα αυτό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης απέρριψε έτσι και αλλιώς και τα διεθνή επίπεδα για την συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Γιατί είναι τόσο επιφυλακτική απέναντι στο blending η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι χρήσιμο ένα τέτοιο μέσο για τις λεγόμενες χώρες ενδιαμέσου, μεσαίου οικονομικού επίπεδου. Είναι ένα, ένα, μια εξαιρετική ιδέα που θα βοηθήσει τις χώρες αυτές να χρησιμοποιήσουν με τη μορφή μόχλευσης τη συμμετοχή του δημοσίου. Πάντως και για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, για την Αφρική βλέπουμε ότι δεν πετυχαίνουν τους στόχους ε, της αύξησης ε, που προβλέφθηκε για την Αφρική. Ε, μήπως εδώ λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και να εξαντλήσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Γιατί οι χώρες αυτές ε, χρειάζονται όλο και περισσότερο τα, ε, τις διαθέσιμες πιστώσεις. Και τέλος άκουσα ότι <laughs> άκουσα και τη φωνή κάποιων Σκανδιναβών στις ε, ομιλίες που προηγήθηκαν την Παρασκευή στο Όσλο θα υπάρξει μια συνάντηση των ε, εκκλησιαστικών οργανώσεων βοήθειας και θα τεθεί το ερώτημα φτάνουμε στο τέλος της, του, στο τέλος σε βάση περιπτώσει του σκανδιναβικού παραδείγματος, της σκανδιναβικής πρωτοπορίας, γιατί μιλάμε για μείωση της χρηματοδότησης, όχι μείωση απλά κατάρρευσης της χρηματοδότησης κατά 50%. Βλέπετε ότι πολλές οργανώσεις από τον επόμενο χρόνο δεν θα μπορούν παρά να εξυπηρετούν σε ελάχιστη βάση τους στόχους τους. Η Νορβηγία αποφάσισε τώρα το 60% της αναπτυξιακής της βοήθεια θα δοθεί στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης αλλά δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι σωστό και αν ισχύει για τη Σουηδία και τους Δανούς. Θα ήθελα οι δύο, δαν, οι δύο ομιλητές. Φτάνουμε λοιπόν στην αρχή του τέλους αυτής της ε, σκανδιναβικής πρωτοποριακής εμπλοκής και νομίζω ότι συνδυαστικά η σκανδιναβική βοήθεια έφτανε το 50% των Ηνωμένων Πολιτειών, της αντίστοιχης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντικό ποσοστό αυτό. Πρέπει να το συζητήσουμε και είναι υπόλογη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μέρος και να μας δώσει στοιχεία για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πιο ενδιαφέρον στην έκθεση είναι οι προκλήσεις και το τι έχουμε ενώπιόν μας. Και υπάρχει, ξέρετε, στα γερμανικά μια έκφραση που λέει ότι το αντίθετο του καλού είναι η καλή πρόθεση. Και αυτό φαίνεται με το ότι στο παρελθόν στην αναπτυξιακή πολιτική και τα κρατημέλη αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν μεν καλές προθέσεις, είχαν διαθέσει κονδύλια για διαφορά έργα κτλ. Και είχαν την εντύπωση ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έτσι. Διοχετεύοντα λοιπόν κονδύλια αναπτυξιακή βοήθεια κάπου στην Αφρική, κάπου στην ε, Κεντρική και Νότια Αμερική, όμως πιστεύω πως αυτού του είδου η πολιτική έχει φτάσει στα όρια της, έχει φτάσει στο τέλος. Έχει αλλάξει και ο κόσμος το κάτω-κάτω. Και εάν ισχύει αυτό που διάβασα πρόσφατα, ότι δηλαδή πριν από 30 χρόνια οι ροέ ε, κονδυλίων στι αναπτυσσόμενε χώρε ήταν, αποτελούσαν το 70% του ΑΕΠ και ότι τώρα είναι μόνο το 7% ε, δημιουργεί τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις. Πάρα πολλές από αυτές τις χώρες δεν είναι φτωχές καθ' αυτές. Ο κόσμος είναι φτωχός εκεί. Τα κράτη όμως, ε, οι περιφέρειες, οι κυβερνήσεις είναι πλούσιες. Το έδαφος είναι πλούσιο, το υπέδαφος είναι πλούσιο σε πρώτες ύλες, δεν είναι λοιπόν φτωχές χώρες, έχουν φτωχούς ανθρώπους. Και το θέμα είναι που πηγαίνει η αναπτυξιακή βοήθεια. Ο πλούτος δηλαδή που έχουν αυτές οι χώρες ε, φαίνεται πως ε, δεν ωφελεί καθόλου τους κατοίκους τους. Και χρειάζεται μία αλλαγή στο αφήγημα της αναπτυξιακής βοήθειας, πιστεύω πρέπει πλέον να σταματήσει να γίνεται τόσο πολύ λόγος για αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά στο πώς θα είμαστε περισσότερο δίκαιοι σε αυτήν την αναπτυξιακή βοήθεια, πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτόν τον ολόνα και περισσότερο δικτυωμένο κόσμο. Επίσης μην ξεχνάμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μάλλον προέρχεται περισσότερο από δημόσιους πόρους από τον προϋπολογισμό του κράτους, από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ιδιαίτερα τώρα σε αυτές ε, τις ε, εποχές κρίσης που ζούμε είναι ολοένα και πιο δύσκολο να τραβήξουμε κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και μάλιστα διάβασα πρόσφατα ότι η Apple για παράδειγμα είχε 17 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη το περασμένο έτος. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο είναι ίσο με τις επερικοπές που έγιναν στον δημόσιο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δηλαδή διαπραγματευόμαστε το, ε, για το πόσο θα κόψουμε από τους κρατικούς περιπολογισμούς και βλέπουμε ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν τόσα υψηλά κέρδη. Επιχειρήσεις μάλιστα και όχι όπως η Apple και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες αυτές χώρες, αποψηλώνουν τα δάση τους, εξαντλούν όλους τους ε, φυσικούς πόρους που διαθέτουν χωρίς να δίνουν τίποτα πίσω. Εμείς πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι προκλήσεις έχουμε ενώπιόν μας και πώς θα καταπολεμήσουμε αυτές τις ανισότητες, τη φτώχεια που μαστίζει τον ε, πληθυσμό εκεί. Και δεν αρκεί λοιπόν να δίνουμε απλά οικονομική αναπτυξιακή βοήθεια για να γίνουν όλα αυτά. Χρειάζεται να υπάρξει μια θεμελιώδης αλλαγή στην αναπτυξιακή μας πολιτική. και είναι μια πολύ υπεύθυνη θέση αυτή του υπεύθυνου ανάπτυξης. Από την άλλη πρέπει να αναγνωρίσουμε επιτέλους τη διασύνδεση της αναπτυξιακής πολιτικής με την εμπορική πολιτική, με την οικονομική πολιτική. Και αυτό έχει άμεση σχέση με το πώς εμείς πρέπει να αντιμετωπίζουμε πλέον τις εμπορικές μας και τις οικονομικές μας σχέσεις με αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις οποίες στέλνουμε αναπτυξιακή βοήθεια. Οι προκλήσεις δηλαδή για μένα είναι αλλού και όχι εκεί που αναφέρεται. Μάλιστα. Είχαμε πιο πολλά θέματα ετέθησαν και παρατηρήσεις έγιναν και ερωτήματα προς τους ε, ομιλητές. Θα δώσω αμέσως το λόγο στο πάνελ για να απαντήσει γιατί έχουμε και τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και την COP21. Ένας στόχος, στον οποίο δεν τα έχουμε καταφέρει και τόσο καλά, είναι η άσκηση της χρηματοδότησης προς τις λιγότερο αναπτυσμένες χώρες. Και το ερώτημα μου είναι, πώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση που να αφορά μόνο τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρε για να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, πόσο καλά λειτουργεί το blending. Ιδίω όταν λέμε ότι ε, ακολουθούμε μια νέα προσέγγιση που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ή στα φορολογικά έσοδα, πόσο αυτά τα νέα, η νέα προσέγγιση, αυτά τα μέτρα ωφελούν τις ε, λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες σε περιοχές όπως η λοιπόν Σαχάρη Αφρική όπου γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι απογοητευτική. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς σε αυτές τις χώρες ε, τι αποτελέσματα έχει η πολιτική μας. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος του ΩΣΑ πρέπει να μετράμε περισσότερο τον αντίκτυπο, τα αποτελέσματα και όχι τόσο τις διαδικασίες ή τα μέτρα που λαμβάνουμε. Γιατί πιθανώ κάποια από τα μέτρα που να λαμβάνουμε να βοηθάνε ιδιαίτερα τι χώρε του μέσου εισοδήματο και όχι τόσο τι λιγότερο αναπτυγμένε. Βεβαίω γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που παίζουν κάποιο ρόλο, όπω οι εμπόλεμε συγκρούσει, αλλά μήπω καλύτερα θα ήταν ε, η αξιολόγηση και οι εκθέσει μα να βασίζονται, ε, να, να δομούνται με βάση τα αποτελέσματα και όχι τόσο τι διαδικασίε μα. Θα δώσω το λόγο στου ε, ομιλητέ του πάνελ με την αντίστροφη σειρά. Α αρχίσουμε τον εκπρόσωπο του ΩΣΑ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής για τα εξαιρετικά σχόλια που έκαναν και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς ποιοι θα είναι οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για τους ε, βιώσιμους στόχους. Φοβάμαι όμως ότι θα είναι πολύ συντηρητικοί και δεν θα μας βοηθήσουν να εστιάσουμε στα αποτελέσματα, όπως είπα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δείκτες δηλαδή του αντικτύπου. Ίσως να μην ε, χρειάζεται να μετράμε και τους 300 που έχουν προταθεί. Ίσως ορισμένοι από αυτούς να είναι οι πιο σημαντικοί εκείνοι που πραγματικά ε, μετρούν την πρόοδο ε, στις διάφορες χώρες επιτόπου. μου αρέσει η παρατήρηση που έγινε για το εάν τελικά θα πρέπει να είμαστε να λογοδοτούμε όσον αφορά την υλοποίηση του ε, στόχου 17 ή αν θα πρέπει να λογοδοτούμε για την ε, υλοποίηση και των 17 στόχων. Πραγματικά εγώ πιστεύω το δεύτερο, γιατί μόνο τότε θα καταφέρουμε να μετρήσουμε αν πραγματικά υπάρχει πρόοδος, διαφορετικά θα παραμείνουμε σε αυτό που κάναμε ως τώρα, μια αξιολόγηση των διαδικασιών. Ε, Παλαιότερα ήμουν και γενικό διευθυντή τη NORAD, τη ε, Νορβηγική Υπηρεσία Αναπτυξιακή Συνεργασία. Γνωρίζω λοιπόν τα θέματα που θέσατε, ε, κυρία Χούταλα, και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσω και μια ανακοίνωση σε σχέση με ε, την σκανδιναβική αναπτυξιακή βοήθεια. Πράγματι έχετε δίκιο ότι αλλάζουν τα πράγματα στι σκανδιναβικέ χώρε δεν πιστεύω ότι βρίσκονταν και τόσο πολύ στην πρωτοπορία οι σκανδιναβικέ χώρες κατά το παρελθόν. Πράγματι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια από τις σκανδιναβικέ χώρες ήταν υψηλή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο την ε, αποστέλαμε στις ε, ε, χώρες που, την, που δεν ήταν και τόσο πρωτοποριακός. Πράγματι με ανησυχούν οι αλλαγές που γίνονται στη Φιλανδία και στη Δανία. Ωστόσο, η ανακατονομή του προπολογισμού που παρατηρούμε στην Νορβηγία είναι εύλογη, είναι κάτι που συμβαίνει διαρκώς, το ίδιο και για την Σουηδία. Το ζήτημα όμω είναι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ΟΣΑ και για όλους. Αν αρχίσουμε να μετράμε την, τα χρήματα που δαπανούνται για την αντιμετώπιση της, προ, της προσφυγικής κρίσης ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, ε, θα έχουμε μια πλασματική αύξηση των ποσών που φαίνεται να δίνουμε για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να προσπαθήσει κανείς να παρέμβει στις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες παρά να ξοδεύει χρήματα για να υποδέχεται τους πρόσφυγες από τις χώρες αυτές. Και άλλα πολλά θα ήθελα να πω, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μια επόμενη ομιλήτρια. Βέβαια, είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε δείκτε για του ε, στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι κάτι το διαφορετικό. Ε, το, η έκθεση για το SDG, εφόσον δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση, δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δεύτερον, σχετικά με την φοροεισπρακτική ικανότητα των μηχανισμών στις υποανάπτυξη χώρες. Με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό. Είδαμε ότι το Δέλτα Ταφ και η Παγκόσμια Τράπεζα πιέζει προς τις ε, χώρες αυτές ε, να φορολογήσουν ε, τους καταναλωτές, τις μητέρες που πηγαίνουν στα καταστήματα να αγοράσουν τρόφιμα για την οικογένειά τους. Οι φτωχοί λοιπόν πληρώνουν φόρους στις χώρες αυτές, οι πλούσιοι όμως και οι επιχειρήσεις όχι. Υπάρχουν ορισμένες χώρες μέλη που δεν είναι και ιδιαίτερα επίμονες σε σχέση με το να πληρώνουν φόρους ε, τα, οι επιχειρήσεις τους. Και οι ίδιες αυτές χώρες στέλνουν κυβερνητικούς εκπροσώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες να βοηθήσουν την σφοροεισπρακτική τους ε, ε, ικανότητα. υπάρχουν ένα παράδειγμα με αυτούς τους ε, τους ελεγκτές τους, ε, της φορολογίας οι οποίοι ελέγχονται από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε την πρωτοβουλία αυτή να την ελέγξουμε, διότι ας μη θεωρήσουμε ότι κάθε μορφή βοήθειας για την ανάπτυξη των φορολογικών συστημάτων θα έχει σώνει και καλά ένα happy end. Το τελευταίο λεπτό που έχω στη διάθεσή μου για τη Δανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Πράγματι υπήρχε μια ειδική, αν θέλετε, σκανδιναβική διάσταση στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόντουσαν με τις αναπτυσσόμενες χώρες και στον τρόπο που βοηθούσαν τις χώρες αυτές να βοηθήσουν τον εαυτό. Δυστυχώς όμως αυτό έχει αρχίσει και καταραίει. Ε, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει κανένας τις χώρες αυτές να πάρουν ε, μια θέση στα διεθνή φόρα. Αυτό δεν κοστίζει τίποτα. Από την άλλη υπάρχει και αναπτυξιακή βοήθεια η οποία δεν εξαφανίζεται αλλά ανακατευθύνεται. Ας πούμε οι στόχοι και τα χρήματα για τους στόχους της Δανίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη και των δανέζικων επιχειρήσεων. Γιατί, γιατί οι δανέζικες επιχειρήσεις είναι η καλύτερη περίπτωση ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, ή μήπως ε, έχουμε δημιουργήσει εδώ κάποιο πεδίο σύγχυσης. Ξέρουμε τι γίνεται με τις αιωλικές από τη Δανία στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά αυτό δεν έχει κάτι να κάνει ιδιαίτερο με την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας για τα σχόλιά σας, τέσσερα σύντομα σημεία. Καταρχάς, το θέμα των εμβασμάτων. Αυτό είναι κάτι που τέθηκε και από την κυρία Σλάινα έχει υπάρξει συζήτηση για τη μείωση του κόστους και αυτό αμφισβητήθηκε βέβαια για τον ρόλο μακροοικονομικά που πρέπει που να παίζουν αυτές οι διαδικασίες των εμβασμάτων και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούνται κυρίως όχι τόσο για εσωτερικές επενδύσεις αλλά για την αύξηση της κατανάλωσης. Η συζήτηση λοιπόν είναι σχετικά περίπλοκη εδώ και δεν αφορά αποκλειστικά τη μείωση του κόστους της συναλλαγής. Δεύτερον, θα ήθελα εδώ να επαναλάβω την δήλωση των συναδέλφων για την αύξηση ακριβώς ε, των ικανοτήτων των φορολογικών των διαφόρων χωρών. Κάποια θετικά σημεία εδώ μπορεί να υπάρξουν. Νομίζω όμως ότι το βασικό θέμα στο οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεισφέρει ε, είναι να χρησιμοποιήσει φυσικά τους εσωτερικούς πόρους μέσω συγκεκριμένων πολιτικών, συνεκτικών πολιτικών και η πρωτοβουλία αυτή η φορολογική ε, την οποία πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνουν αφορά ακριβώς τη συνεκτικότητα ε, και είναι πολιτικά θα έλεγα ένα τέτοιο θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα τρίτο σημείο για την σκανδιναβική εξαίρεση. Ακόμα και στην χρήση των ODA για διαφορετικούς στόχους δεν είναι κάποια εξαίρεση, έχει συμβεί στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες. Όχι μόνο για το κόστος κάλυψης των προσφύγων, αλλά και για την χρήση ε, των μέσων αυτών για την προώθηση των εθνικών πολιτικών. Αυτό είναι θεμητό θα έλεγα όχι όμως για την ανάπτυξη, δεν βοηθάει άμεσα την ανάπτυξη. Και ένα τελευταίο θέμα ε, για, το, για την αναγνώριση ακριβώς της επίσημης συνολικής βοήθειας μεμονωμένα από χώρες. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην προχωρήσουμε στην απίσχναση των ODA επιδιώκοντας βέβαια κάποιους άλλους θεμητούς στόχους. Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να πάνε στις φτωχές χώρες για τους φτωχούς πληθυσμούς τους να χρησιμοποιηθούν για άλλο στόχο. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να απαντήσω επαρκώ σε όλε τι ερωτήσει και τα σχόλια εντό τριών λεπτών, αλλά θα προσπαθήσω. Καταρχά, η έκθεση λογοδοσία. Όταν την καταρτήσαμε ή είχαμε ένα άλλο καθεστώς και θεωρούσαμε πως δεν επαρκούσαν, για παράδειγμα, οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας και η εξετασή τους κάθε πέντε χρόνια. Θέλαμε να εφαρμοστεί η λογοδοσία και εννοώ να εφαρμοστεί και στα θεσμικά όργανα και στα κρατημέλη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάστηκε να ασκήσουμε πίεση στα διάφορα κρατημέλη έτσι ώστε να προχωρήσουν και να αναγκαστούν να συζητήσουν το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα σχετικά με την εφαρμογή της ε, Συμφωνίας του Μοντερέι. Αυτό θα αλλάξει. Θα υπάρχει ένα σύστημα λογοδοσίας σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και για τους βιώσιμους ε, στόχους της ανάπτυξης και για την έκθεση. Εμείς Θέλουμε να φροντίσουμε να υπάρχει τέτοια οργάνωση έτσι ώστε να μην εξετάζονται τα δύο αυτά ε, πράγματα ξεχωριστά. Πρέπει να επιφέρουμε τη συνοχή. Και πιστεύω πως ε, και η Αντίσαμπεμπα και η Νέα Υόρκη είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έξεσή μας. Και πιστεύουμε πως ε, μπορούμε μαθαίνοντας από τα όσα έγιναν στην Αντίσαμπέμπα και στη Νέα Υόρκη να αλλάξουμε το αφήγημα. Να αλλάξουμε το αφήγημα και να καταστήσουμε υπεύθυνους όλους. Υπεύθυνους για τα έργα τους, για τις πράξεις τους, για τις υποσχέσεις τους. Δηλαδή ότι εμείς αναλαμβάνουμε να κάνουμε, να αναλαμβάνουμε και τη σχετική ευθύνη. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω πως ε, σε σχέση με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και τις δεσμεύσεις μας πέρα από αυτή, βέβαια χρειαζόμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας θέλουμε να επικοινωνήσετε με τα εθνικά σας κοινοβούλια και να το απιέσετε, γιατί χρειάζεται πίεση. Και επίσης σχετικά με τις ε, βόρειες χώρες και την Ορβηγία. Πράγματι υπήρξε κάποια μείωση, δηλαδή η Δανία έπεσε στο 0,7 αντί να το ξεπεράσει και κάποιες άλλες χώρες, η Γερμανία νομίζω αύξησε την αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει όμως ε, να σταθούμε στις χώρες οι οποίες είτε αύξησαν την αναπτυξιακή βοήθεια είτε θα την αυξήσουν στο μέλλον. Ας δούμε δηλαδή το σύνολο της Ευρώπης. Τώρα, το φορολογικό σύστημα. Σίγουρα όσα και οι g κάνουν καλή δουλειά. Υπάρχει και μια επιτροπή φορολογικών υποθέσεων στα Ηνωμένα Έθνη. Βέβαια υπάρχουν συνάδελφοί μου που είναι πολύ πιο αρμόδιοι και πολύ καλύτερα καταρτισμένοι από εμένα για να σας ε, εξηγήσουν τα φορολογικά ζητήματα και το τι κάνουμε εμείς για να στηρίξουμε το φορολογικό σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύουμε όμως πως αυτός ε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Τώρα, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως μπορούμε να επανεξετάσουμε με περισσότερη προσοχή κάποια από τα ζητήματα που θίξατε και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Εντάξει, όσο για το φυλάδιο που λάβατε, θα φροντίσω να λάβατε και, το, και την έγχρωμη εκτύπωση, έτσι ώστε να δείτε καλύτερα τα γραφήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέραν αυτών, να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα και μετά, βασισμένοι σε αυτά, να προσαρμόσουμε και τις λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό πιστεύω ήταν πολύ καλό να, που το ακούσαμε. Θέλουμε να δούμε πώς προχωράτε. Και μπορούμε νομίζω να ζητήσουμε και από τους συντονιστές να διοργανώσουν μια ανταλλαγή απόψεων για να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται και με εσά και με τον ΟΣΑ και με τους άλλους φορείς. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω και τους τέσσερις ε, προσκεκλημένους για την εξαιρετική παρουσία Τώρα θα αλλάξει το πάνελ και θα ήθελα να προσκαλέσω στο Προεδρείο τους προσκεκλημένους για την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Μακουέιντ βλέπω είναι πάλι εδώ και του λείψαμε από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Τεγκόλφι βλέπω είναι εδώ η κυρία Κουίν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 Περνάμε λοιπόν ευθύ αμέσω στην παρουσίαση. Um, Καθίστε παρακαλώ, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά η προηγούμενη συζήτηση κράτησε λίγο περισσότερο. Επόμενο θέμα μας είναι η διάσκεψη στο Παρίσι, σε δυόμιση μόλις εβδομάδες. Ήμουν στην διάσκεψη της Κοπενχάγης και δούλεψα μεταξύ άλλων και για τον περιβαλλοντικό νόμο, την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ένα από τα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν στην Κοπενχάγη είναι πώς οι αναπτυσσόμενες χώρε θα υποφεληθούν από μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Και για να οδηγηθούμε βέβαια σε μια παγκόσμια συμφωνία πρέπει να έχουμε κατά νου και τις αναπτυσσόμενες χώρε. Είναι οι δύο πλευρέ δηλαδή του ίδιου νομίσματος. Έχω την κυρία Κουίν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω εκπρόσωπο από την ε, ε, ΓΔ ο κ. Μακλίν από το Climate Action Network. Η Τατιάνα Νάμπης από το ΒΒΕΒ. Και το ΒΒΕΒ συμμεταχεί ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Θα έχετε πέντε λεπτά χρόνο καθένα. Θα αρχίσουμε από την κυρία Κουίν, αναπληρώτρια τμήματάρχης για ε, θέματα κλιματικής αλλαγής και χρηματοδότησης. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να αρχίσω τονίζοντας ότι το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ έχει ψηφίσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το κλίμα και τη χρηματοδότηση σήμερα. Πιστεύω πως οι γενικές γραμμές είναι αρκετά καλά. Υπάρχει μια δέσμευση για αύξηση της χρηματοδότησης για, την, για το κλίμα τα επόμενα χρόνια. Και επίσης θα γίνει ένας απολογισμός ε, του πού βρισκόμαστε. 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύτηκαν για την ε, κλιματική αλλαγή το 2015. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου επίσης καλωσόρισαν την ε, προσφατή έκθεση του ΩΣΑ για την πρόοδο προς τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2020. 100 δισεκατομμύρια για το κλίμα. Τώρα έχουμε φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, το Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε να φτάσουμε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Επίσης δημιουργείται το πλαίσιο και η διαπραγματευτική εντολή για την ε, διάσκεψη στο Παρίσι για τη συνέχεια της ε, συμφωνίας μετά το 2020. Επίκεντρο είναι οι πιο φτωχές, πιο ευάλωτες χώρες και η προσαρμογή στην χρηματοδότηση. Επίσης, στάλησαν ισχυρά μηνύματα προς τον ιδιωτικό τομέα να μειώσει τις εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου και να συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή. Και επίσης, να βοηθήσει στην κατάρτιση σχεδίων, ε, ρυθμιστικών πλαισίων και μέσων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν ε, πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει ένα σύστημα τιμολόγησης, ένα σύστημα φορολόγησης ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και το πιο σημαντικό πιστεύω από όλα αυτά είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης έχουμε το Ταμείο Προσαρμογής, το οποίο έχουμε κατά 50% ε, εξοπλίσει με κονδύλια. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020 να αυξήσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το κλίμα και για το περιβάλλον. Στην ουσία θα προσπαθήσουμε να διπλασιάσουμε τα κονδύλια που διαθέτουμε έτσι ώστε να φτάσουμε τους στόχους του 2020. Τώρα, αρκετά κράτη-μέλη επίσης δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις συνεισφορές τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά είναι λίγοι σε το τι θέλαμε μέχρι τώρα. Τώρα, η Συμφωνία του Παρισιού πρέπει να δημιουργήσει μία παγκόσμια ε, νομικά δεσμευτική συμφωνία που θα διακρίνεται από διαφάνεια, από λογοδοσία και που θα απαντά στην ανάγκη πιο φιλόδοξων στόχων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, ανάληψη, αναλήψη υποχρεώσεων από πάνω από 130 χώρες για την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και θα συνεχίσουμε αυτές τις φιλόδοξες δεσμεύσεις. Θα γίνουμε ακόμα πιο φιλόδοξοι. Είναι δύσκολη όμως η διαπραγμάτευση για την χρηματοδότηση της ε, κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες ε, ζητούν χρηματοδότηση, εμείς δεν θέλουμε πως είναι τόσο βαθύ το χάσμα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει διευρυνθεί η βάση των δωρητών, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν αλλάξει οι κατευθύνσει των ε, χρηματοδοτικών ροών, ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο για την κλιματική αλλαγή. Έτσι λοιπόν δεν στεκόμαστε μόνο στις ε, αναπτυγμένες ε, παραδοσιακά χώρες, αλλά έχουμε επεκταθεί και στις αναπτυσσόμενες χώρες για την χρηματοδότηση του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τώρα την κλίμακα και τους πόρους, εδώ βλέπουμε πως υπάρχει ανάγκη για μια μεγάλη μετάβαση προς μια οικονομία ανεξάρτητη από το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό φυσικά έχει υψηλό κόστος και τα δημόσια οικονομικά δεν αρκούν να το καλύψουν. Το πιο σημαντικό είναι να κατευθύνουμε σωστά τις επενδύσεις και να συμπεριληφθεί και ο ιδιωτικός τομέας στους επενδυτές. Έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε τις δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις χώρες. Η στάση της Κίνας ίσως αποτελεί εμπόδιο για κάποιους, όμως εμείς δεν έχουμε τέτοια άποψη. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές ε, στην κλίμακα, στην τάξη μεγέθους, δηλαδή οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούν ξεκάθαρες δεσμεύσεις, ποσοτικές δεσμεύσεις, κάτι που είναι μια αντιμετώπιση διαφορετική από εκείνη των ε, αναπτυγμένων χωρών. Επίσης χρειάζεται διαφορετική δυναμική στη χρηματοδότηση, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λεποδοσία, να ξέρουμε τι δίνουμε και πού το δίνουμε. Και αυτό συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από κλιματικούς στόχους, από στρατηγική ανάπτυξη, από στήριξη των προσπαθειών, από προσπάθειες για αύξηση της διεθνούς χρηματοδότησης. Καθώς και από διαφάνεια των οικονομικών. Είναι δύσκολο το ζήτημα και πιστεύω πως η επίλυσή του θα είναι και αυτή δύσκολη. Θα είναι το τελευταίο ίσως δύσκολο κομμάτι των διαπραγματεύσεων διότι είναι ένας τομέας όπου ίσως παρατηρούνται οι μεγαλύτερες διαστάσεις απόψεων. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει μια διαφορετική στάση για την χρηματοδότηση για το περιβάλλον και υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις άλλωστε ανάμεσα και στις δυτικέ χώρες. Σίγουρα θα πρέπει να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Αυτά από μένα προς το παρόν. Ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι συνεργάζεστε στενά ε, με την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπό της. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος κάλυψε περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω για τη χρηματοδότηση ε, τη αναπτυξιακή και η χρηματοδότηση της καταπολέμησης τη κλιματική αλλαγή. Αυτά τα δύο είναι οι δύο όψει του ίδιου νομίσματος. Δεν γίνεται να συμβεί το ένα χωρί το άλλο. Πρέπει να καταπολεμηθούν οι ανισότητες οι οικονομικές και να καταπολεμηθεί η φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι και οι πιο βάλλοντες στους κινδύνους που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Γιατί συνήθως οι χώρες αυτές βασίζονται στο τομεί της οικονομίας που εξαρτώνται από τις συνθήκες τις μετεωρολογικές και επίσης επειδή έχουν πολύ λιγότερους πόρους στη διάθεσή τους για να αντιμετωπίζουν τις κλιματικές αλλαγές Επομένως θα πρέπει η ανάπτυξη που προωθούμε στις χώρες αυτές να είναι ε, να μην, να μην δημιουργεί προβλήματα κλιματικά και να μπορεί να αντισταθεί στην κλιματική αλλαγή ήδη από την αρχή. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα που κομίζουμε στο Παρίσι και πιστεύω ότι η αναπτυξιακοί στόχοι, οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι μας δίνουν ένα καλύτερο περιβάλλον γιατί επιτυγχάνοντας έναν από αυτούς, διευκολύνεται η επίτευξη των άλλων. Στη Νέα Υόρκη αναγνωρίστηκε και ετέθη ένας ξεχωριστός στόχος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, το οποίο δείχνει, ε, δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η διεθνή κοινότητα αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της ε, αντιμετώπισης τη κλιματικής αλλαγής, αλλά και ταυτόχρονα ότι δεν μπορεί αυτή η αντιμετώπιση της αλλαγή του κλίματο να γίνει ε, χωριστά και αποσπασμένα από του υπόλοιπου αναπτυξιακούς στόχους. Αυτό ε, φαίνεται σε πολλούς τομείς, για παράδειγμα στην αγροτική παραγωγή, στη Γεωργία. από τι επισκέψει μου σε χώρε όπω η Ουγγάντα γνωρίζω ότι η έρευνα που γίνεται για νέες μεθόδους ε, αγροτικής ανάπτυξης είναι ήδη από μόνη της μια ε, πρωτοβουλία που θα βοηθάει στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη είναι ένας από τους κυριότερους χρηματοδότες των προσπαθειών των χωρών αυτών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το 2014 είπατε ότι αυξήθηκε σε σχέση με το 2013, αλλά θα πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοδότηση. Και θα, από όλα τα πιθανά χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την, το DCI για την επίτευξη του στόχου μέσα στο 2020. Θέλουμε να ξεπεράσουμε στον στόχο του 20%. Αλλά επίσης, το πλαίσιο των SDG με τους δείκτες μας υπαγορεύουν τι θα έπρεπε να κάνουμε κάθε μέρα, καθημερινά. Το οποίο σημαίνει, εάν χρηματοδοτήσω το ΑΒ έργο, πόσοι άνθρωποι θα ωφεληθούν πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει την αλλαγή του κλίματος. Εμείς είχαμε βασιστεί σε ένα σύστημα το οποίο ε, που βασιζόταν στις δεσμεύσεις και μετά στην πληρωμή με βάση τις δεσμεύσεις. Και τώρα προσπαθούν όλοι να, να, να αλλάξουν την προσέγγιση τους. Στην Κοπεχάγη η προσέγγιση ήταν είτε θα τα συμφωνήσουμε όλα, είτε θα συμφωνήσουμε τίποτα. Και τελικά δεν συμφωνήσαμε σε τίποτα. Στο Παρίσι ακολουθείται μια διαφορετική προσέγγιση. Θα συμφωνήσουμε σε ένα ελάχιστο μέσο όρο τώρα, σε ένα ελάχιστο κοινό και κάθε τρία χρόνια θα υπάρξει μια αναθεώρηση. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί γνωρίζουμε ότι οι επιστημονικές ε, εκτιμήσεις διαφέρουν, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από κάτι αυτή τη στιγμή. Χωρίς να πω τώρα σε συγκεκριμένα στοιχεία που ίσως το συνάδελφος από τη ΒΒΕΦ ή από άλλες κυβερνητικέ οργανώσεις για το περιβάλλον θα μπορούσαν να μας δώσουν καλύτερα. Το ζήτημα επίση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ποια είναι η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα σε, αυτού, σε αυτή τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή είναι μεγάλη σήμερα, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μα αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η χρηματοδότηση θα προέρχεται κυρίως από τους κρατικούς πόρους, από τη δημόσια χρηματοδότηση. Θα πρέπει να έρθει κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως θα πρέπει να βρούμε τρόπους να κινητοποιήσουμε, να ενθαρρύνουμε τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα συζητά ποιο θα είναι ο ρόλο του ιδιωτικού τομέα επί τη βάση τη ανακοίνωση τη Επιτροπή. Συζητείται ακόμα στο Συμβούλιο, συζητείται και στο Κοινοβούλιο. Αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο πολιτική. Χωρί αυτό δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει, να συνεισφέρει του επιπλέον πόρου που μα λείπουν ε, από τον ιδιωτικό τομέα θα έρθουν αυτοί οι πόροι που μας λείπουν. Δεν μπορούν να καλυφθούν από, τον, από τους δημόσιους πόρους. ο στόχος για τον εξηλεκτρισμό. Είναι 100% συνδεόμενος με την αντιμετωπίση της κλιματικής, γιατί θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές ε, να έχουν πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια. Ο στόχος που αφορά στις βέλτιστες πρακτικές τη γεωργία έχει σχέση με την ε, ενθάρρυνση περισσότερων ε, ιδιωτικών επενδύσεων για ε, περιβαλλοντικά βιώσιμους τρόπους αγροτικής ανάπτυξης. Πολλά κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισέφεραν έως τώρα στην προετοιμασία μας, της παρουσίας μας στο Παρίσι, προσπαθούμε να διοργανώσουμε και διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις και πιστεύω ότι το σημαντικότερο θα είναι οι αντιπροσωπείες μας να επιμείνουν στο στόχο του 20% και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό έτσι ώστε ο σχεδιασμός που θα γίνει να ταιριάζει με αυτόν τον στόχο του 20%. Και ελπίζοντας ότι κατά την υλοποίηση θα το ξεπεράσουμε το 20% ακόμα περισσότερο. Σα ευχαριστώ να ακούσαμε του δύο εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα θα δώσω του λόγου στου εκπροσώπου των δύο μη οργανώσεων. Ξεκινώντα από τη σημασία για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Μπορείτε να μα δώσετε κάποιε περισσότερε πληροφορίε για την οργάνωση που εκπροσωπείτε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλο και περισσότερο βλέπουμε να δημιουργούνται συνέργειες ε, λόγω ακριβώς των κοινών ανησυχιών που έχουμε εμείς λόγω των ε, κλιματολογικών συνεπειών. Υπάρχουν ε, λοιπόν αρκετές μικιό που ασχολούνται με τα θέματα της αηφορίας αλλά ειδικότερα με τα θέματα των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών και με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται. Και το θέμα επίσης της χρηματοδότησης των δράσεων στον τομέα των κλιματολογικών. Θα ήθελα να σας μεταφέρω ποιες είναι οι ανησυχίες των ΜΚΟ αλλά και ποιες είναι οι ανησυχίες των αναπτυσσομένων χωρών. Ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από το ΕΚΟΦΗΝ ε, σήμερα αν παρουσίαζα τις θέσεις αυτές στους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών θα ένιωθαν μια τρομερή δυστημία για την έλλειψη φιλοδοξίας η οποία υπάρχει και εγώ μίλησα με εκπροσώπους του Νεπάλ, της Τανζανίας, της Ζάμπια και το θέμα της χρηματοδότησης τους στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού είναι σημαντικότατο για αυτές τις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής, είναι παραδοσιακός σύμμαχος των αναπτυσσομένων χωρών. Δεν μπορώ να προκαταλάβω εγώ τα συμπεράσματα αυτά, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν είχαν την δυνατότητα οι αναπτυσσόμενες χώρες να εκφραστούν, θα καταδίκαζαν αυτή την έλλειψη φιλοδοξίας και από πλευρά των Υπουργών Οικονομικών και από πλευρά των ηγετών των κρατών και των κυβερνήσεων υπάρχει μια πλήρης θα έλεγα έλλειψη βελτίωσης της κατάστασης ακόμα και στα πλαίσια της προετοιμασίας για το επερχόμενο ΚΑΠ21. Ε, τα θέματα της χρηματοδότησης πριν από το 2020 ε, θα τα θέσει η Τατιάνα, αλλά νομίζω ότι εδώ σκιάζεται το τι θα γίνει μετά τη χρημα... για την χρηματοδότηση μετά το 2020 σε σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές και πώς θα επιδιώξουμε κάποιες αλλαγές για την απομάκρυνση από τη χρήση του άνθρακα. Νομίζω ότι θα θέλαμε ένα αποτέλεσμα σαφές, απτό και προβλέψιμο, έτσι όπως χώρες των Νεπάλ, η Τανζανία, η Ζάμπια, να προγραμματίσουν και για τα προγράμματα προσαρμογής και για τα προγράμματα μετρίασης των συνεπειών, να μπορούν να υπολογίσουν στη βοήθεια των δωρητριών χωρών και να αναπτύσσουν τις δικές τους ικανότητες. Από ό,τι φαίνεται όμως οι αναπτυγμένες χώρες στην ουσία αυτό το οποίο λέγουν είναι ότι εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε ενώ μπορούν να κάνουν περισσότερα και βραχυπρόθεσμα τα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ δεν καλύπτουν την ανησυχία η οποία υπάρχει ότι θα πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και μετά το 2020. Έχει σημασία λοιπόν να στραφούμε στο μέλλον, θα υπάρξουν πάρα πολλές δυσκολίες και δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη. Σε σχέση με το λεγόμενο mainstreaming, τίθεται το θέμα της προσαρμογής και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της στον τρίτο κόσμο θα μπορέσουν να αυξήσουν την αντοχή τους στις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών και να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα σε ε, χώρες ε, που τα έχουν ανάγκη. Ε, δεν θα πρέπει να εμείνουμε ιδιαίτερα υπερβολικά θα έλεγα σε σχέση με την μετρίαση των συνεπειών, κυρίως όμως σε σχέση με τα προγράμματα προσαρμογής και κυρίως σε σχέση με την χρηματοδότηση των προγραμμάτων προσαρμογής. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των αναπτυσσομένων χωρών, δεν είναι πρόβλημα αυτό για μας, αλλά δεν βλέπουμε να λέγεται πουθενά το τι θα γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο θα δίδεται η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Ποιος θα ελέγχει ακριβώς τον ιδιωτικό τομέα στη συμμετοχή του στην διαχείριση των διεθνών προγραμμάτων. Το θέμα προσαρμογής στις κλιματολογικές αλλαγές δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τον ιδιωτικό τομέα και το ποσοστό απόσβεσης και ο ρυθμός απόσβεσης είναι αρκετά χαμηλότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες από ό,τι στις χώρες μέσων εισόδημάτων. Και τίθεται το θέμα πάντα διαφοροποίησης ανάμεσα στις, ε, στα προγράμματα μετρίασης των συνεπειών από τη μία και στα προγράμματα προσαρμογής από την άλλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν ένας καλός σύμμαχος των αναπτυσσομένων χωρών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, απαιτείται όμως πολιτική ηγεσία και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πλευράς των κρατών μελών. Αυτό είναι ιδιαίτερος κρίσιμο γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα οποία έχουμε ε, ανάγκη στις διεθνείς διαπραγματεύσεις θα πρέπει ακριβώς να ορίσουμε τις θέσεις μας με σωστό τρόπο, να δούμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, μια ολόκληρη διαδικασία σταδιακή αν θέλετε στα πλαίσια των διεθνών διαπραγματεύσεων, τόσο πολύ σημαντική όμως για τις ευαίσθητες χώρες που θα πρέπει να γνωρίζουν τι βοήθεια θα λάβουν στο μέλλον. Και βλέποντας τις συζητήσεις οι οποίες ακούγονται σήμερα, φοβάμαι ότι δεν θα είναι και ιδιαίτερα βέβαιες γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες πριν από τη συνάντηση του COP21 έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τις χώρες ανάπτυξης, με υποανάπτυξη μάλλον χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπολογίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σωστή τους βοήθεια. Η Τατιάνα. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μετά λοιπόν τις ε, πρόσφατες εξελίξεις και τα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ, νομίζω πως ε, θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Καταρχάς υπάρχει ανάγκη για περισσότερη σαφήνεια και διαφάνεια σχετικά με τις ε, ροές των πόρων για την αναπτυξιακή βοήθεια. Από την Κοπεθάκη και πεντά οι χώρες υποσχέθηκαν να διαθέσουν 100 δισεκατομμύρια ε, για την κλιματική αλλαγή και παρότι έχουν, έχουν παρατηρηθεί κάποιες ε, θετικές εξελίξεις υπάρχουν ακόμα ελλείψεις σχετικά με τον ε, τρόπο ελέγχου. Δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα, κοινοί ορισμοί και ορισμένες χώρες παρατηρούν προβλήματα στην λογοδοσία και στην δημιουργία και υλοποίηση έργων. Και αυτό λοιπόν εμείς καλωσορίζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ που ζητούν περισσότερη διαφάνεια και ξεκάθαρους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των ε, χρηματοδοτικών ορών που προορίζονται για το κλίμα. Ακούσατε και εσείς για τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ και για τις ε, διαφορές στον τρόπο ελέγχου στα κράτη-μέλη. Χρειάζονται λοιπόν να ξεπεραστούν τα εμπόδια έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την αναγκαία εμπιστοσύνη. Θα θα ήθελα να αναφερθώ στην ισορροπία ανάμεσα στην χρηματοδότηση για την ε, κλιματική αλλαγή, για την ε, μείωση και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν κονδύλια τα οποία προορίζονται για την ε, προσαρμογή και κάποια άλλα προορίζονται για την μείωση της ε, κλιματικής αλλαγής. Χρειάζεται λοιπόν να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην μείωση και στην προσαρμογή. Χρειάζονται όμω ε, πολλά βήματα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Υπάρχουν ελλείψεις και υπάρχουν, και υπάρχουν προβλήματα που οφείλονται στην παραμέληση των ε, αρμόδιων φορέων να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει περισσότερο τις πιο ευάλωτες ομάδες ε, και τις ε, χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αλλαγής της στάθμης του νερού κτλ. Το κόστος προσαρμογής λοιπόν για τις ε, περιοχές αυτές αυξάνεται και η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις μάλιστα σχετικά με την υποσαχάρια Αφρική. Εκεί εκτιμάται ότι δαπανούν οι κυβερνήσεις αυτές 5 δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή που είναι περισσότερα από όσα λαμβάνουν σαν ε, βοήθεια, σαν αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης χρειάζεται να αλλάξει το βάρος της ε, χρηματοδότησης που αυτή τη στιγμή είναι μόνο στον δημότιο, δημόσιο τομέα. Χρειάζονται λοιπόν ιδιωτικέ επενδύσεις και χρειάζεται πίεση έτσι ώστε οι ιδιωτικές επενδύσεις να γίνουν και σε μη κερδοφόρα έργα για εκείνους, όπως για παράδειγμα ε, τις ε, συνέπειες από τη διάβρωση του εδάφους. Μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για το κλίμα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τώρα βλέπουμε πως παρατηρείται είτε στασιμότητα ή μείωση του κρατικού προϋπολογισμού ε, και σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, αποσπώνται κονδύλια τα οποία διατίθενται για άλλα πολύ σημαντικά προγράμματα, για παράδειγμα για τα καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάτι το οποίο δεν βοηθά. Χρειάζεται φυσικά να αυξηθεί ο προπολογισμό και βλέπουμε ότι κάποιες χώρες όπως για παράδειγμα η Γερμανία έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν ε, τα κονδύλια που διαθέτουν για την αναπτυξιακή βοήθεια, όμως αυτή τη στιγμή χρειάζεται να γίνει πολλά περισσότερα. Έπειτα, χρειάζεται να συγκεντρωθούν κονδύλια και από διάφορες καινοτόμες πηγές, δηλαδή εισοδήματα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, από την ε, πάυση των ε, επιχορηγήσεων για τα ορυκτά καύσιμα και πιστεύω πως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για τη δημιουργία εμπιστοσύνης έτσι ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη διάσκεψη για ε, το Παρίσι. Χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια για τα οικονομικά και τα ποσά που διατίθενται. Χρειάζονται προσπάθειες για προσαρμογή και για μείωση της κλιματικής αλλαγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ έχω τον Ταβοστήρ που έχει ζητήσει τον λόγο και μετά άλλους τρεις συναδέλφους. Παρακαλώ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ομιλητές. Σίγουρα και οι συναδελφοί μου θα μιλήσουν περισσότερο εις βάθος από εγώ για τις ζητήματα αυτά, αλλά έχω ένα ερώτημα για τον πρέσβη Ριντόλφη κάνετε αυτή τη σύγκριση ανάμεσα στην Κοπενχάγη και το Παρίσι. Και όλοι αναφερθήκατε στις προσδοκίες που μπορούμε να έχουμε από το Παρίσι. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Το ερώτημα μου είναι το εξή. Αυτή η τακτική που αποφάσισαμε, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί στο Παρίσι, δηλαδή να εκπροσωπηθούν οι αρχοί κρατών. Αρχικά και, όχι μόνο, και πριν τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Εντάξει, ίσως όλοι να συμφωνούμε ότι δεν είναι δυνατό να επαναληφθεί το φιάσκο της Κοπενχάγης. Αλλά ε, εσείς τι πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει εξαιτίας αυτής της, της προσέγγισης. Ευχαριστούμε. Μετά κύριο Σίλβα και μετά κύριε κυρία Κύριο Σίλβα. Και εγώ στα γρήγορα μια ερώτηση. Θα ήθελα να θέσω στους ομιλητές. που έχει σχέση με την έννοια της προσθετικότητας μια έννοια που την έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε αυτή την Επιτροπή και εις βάθος Δηλαδή, πως η επιπλέον χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του μετριασμό των επιπτώσεων της. Εσείς που έχετε παρακολουθήσει τις παρασκευαστικές εργασίες εν ώψη του COP21, Πιστεύετε ότι το έχουν αντιληφθεί αυτό όλα τα κράτη, ότι συμφωνούν ότι χρειάζονται επιπλέον πόροι και όχι απλώς επανακατανομή των πόρων των υφιστάμενων. Έχουν αντιληφθεί τα κράτη ότι δεν μιλάμε απλώς για μια διαφορετική παρουσίαση του, των χρημάτων που ήδη διαθέτουν και έχουν αντιληφθεί ότι θα χρειαστούν να δώσουν περισσότερα για να επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους. Αν ισχύει μάλιστα μία φορά για του αναπτυξιακού στόχου, ισχύει δέκα φορέ για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, το ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Πώς μπορούμε τελικά να φτάσουμε σε αυτά τα 100 δισεκατομμύρια και να είναι στην πραγματικότητα 100 δισεκατομμύρια. Κύριε θα σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με κάτι που είπατε για τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση λοιπόν για το κλίμα δεν θα πρέπει να προέλθει από την αναπτυξιακή βοήθεια και πρέπει να το τονίσω αυτό. Πιστεύω πως θα είχε μοιραίες επιπτώσεις εάν αντλούσαμε κονδύλια από ένα ε, χώρο ο οποίος χρειάζεται επιγόντως όχι τουλάχιστον τα ίδια αύξηση και όλες. Έπειτα, πιστεύω πως αυτό που χρειάζεται είναι έξυπνες λύσεις, έξυπνες πρακτικές, έτσι ώστε να καταφέρουμε το στόχο μας. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε για τη Γεωργία, έχω τις αμφιβολίες μου. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα, μια, μια πολύ εντατική μέθοδο ε, καλλιέργειας. Τώρα, πρώτες ύλες. Υπάρχει εντατική εξόριξη πρώτων υλών, από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ καταστροφικό αυτό για τη γεωργία. Δηλαδή όταν ας πούμε εξαντλώ το έδαφος από ορισμένα ορυκτά, από ορισμένα μέταλλα, αυτά δεν μπορούν να διοχετευτούν στο χώμα το οποίο θα παράγει με τη σειρά του τρόφιμα. Υπάρχει ο κύκλος του αζότου ας πούμε, τον οποίο μπορείτε να πάρετε ως παράδειγμα. Ε, δεν πρέπει να δώσουμε χρήματα για την γεωργία γενικά και αόριστα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην οικολογική γεωργία, στη βιώσιμη ε, γεωργία και στην ανακύκλωση των ε, υλικών. Αυτό είναι η μόνη λύση και μια οικολογική καλλιέργεια της γης είναι η μόνη λύση έτσι ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αντί λοιπόν να δαπανούμε χρόνο και χρήμα σε πολύπλοκες λύσεις θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε την οικολογική γεωργία. Ε, τώρα πιστεύω πως το χρονικό διάστημα που μας αναφέρατε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Χρειάζεται να επιταχύνουμε την επίτευξη των στόχων μας ε, για να είμαστε και ρεαλιστικοί σχετικά με το τι περιμένουμε. Για τη χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Το ότι η χρηματοδότηση για το κλίμα είναι αιτία διένεξης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δεν είναι κάτι καινούριο δεν έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσει τη Κοπενχάγη για πρόσθετη χρηματοδότηση και αυτό μάλιστα αποτελεί και πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θέλει να υπάρξει πρόοδος προς μια δεσμευτική συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Πριν από κάποια χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια τολμηρή δέσμευση για το έργο, των, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ενέργεια. Και θυμάμαι ακόμα ότι και ο πρόεδρος Μπαρόσο και ο επίτροπος Πίμπαλξ τότε είχαν πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει κατά πολύ έτσι ώστε όσοι δεν έχουν πρόσβαση το ηλεκτρικό ρεύμα για παράδειγμα να μπορέσουν να έχουν και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επομιστεί ένα μεγάλο μέρος του κόστους γι' αυτό. Έχω όμως την αίσθηση πως δεν έχει γίνει τίποτα. Και χρειάζεται λοιπόν χρηματοδότηση, αύξηση της χρηματοδότησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Αν μου πείτε εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη στις δεσμεύσεις. Νομίζω πως αυτές οι δεσμεύσεις που είναι δεσμεύσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο λήφθησαν το 2012. Και τώρα, όπως είπε και η Μαρία Χόιμπουχ, πιστεύω πως η Γεωργία είναι ζωτική σημασία. Εσείς βλέπετε κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να μετατοπιστούμε σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα γεωργίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική. Επίσης, πιστεύω πως πρέπει να είμαστε σε θέση να βρούμε πώς θα μειώσουμε την κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης. Είναι πολύ σπάταλη αυτή η πρακτική και σε ενέργεια και σε παραγωγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εντάξει, δεν λέω να κόψουμε τελείως το κρέας και να τρώμε φύλλα από εδώ και στο εξή όλοι μας, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα. Και εγώ θα ήθελα να πω, να προσθέσω κάτι. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δεσμεύσεις από κάτω προς τα πάνω αντί για το αντίθετο και μην ξεχνάτε ότι αυτή η προσέγγιση top-down, από πάνω προς τα κάτω, είναι επιστημονικά θεμελιωμένη. Υπήρχε λοιπόν κάποια επιστημονική προσέγγιση, κάποια στατιστικά στοιχεία ότι με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το διοξίδιο, οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα βλέπουμε πω ε, την επιστήμη έχει διαδεχτεί η πολιτική και έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και πιστεύω ότι το σκεπτικό του να συνεδριάσουν οι πολιτικοί ηγέτες την πρώτη μέρα του Παρισιού είναι για λόγους στρατηγικής. Για να συζητήσουν το συντομότερο δυνατόν και να έχουν και την προσοχή της κοινή γνώμης τραμμένη προς τα πάνω τους. Και σίγουρα όλοι, κάθε Ευρωπαίος ηγέτης θέλει να δείξει πως είναι ο καλύτερος, ο ισχυρότερος και ο φιλικότερος προς το περιβάλλον. Αλλά κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο, μια και πρέπει να φύγετε. Ευχαριστώ. Ναι, πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα που θα προσκληθούν και την πρώτη μέρα θα ε, συνεδριάσουν οι αρχηγοί κρατών δεν συνηθίζεται με βάση το πρωτόκολλο, έχει δίκιο η Λίντα, αλλά έχει δίκιο επίση που λέει ότι είναι σημαντικό το ότι οι αρχηγοί θα θέσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο από εκεί και πέρα οι τεχνοκράτες και οι υπουργοί θα ε, λειτουργήσουν, θα δράσουν, θα διαπραγματευτούν. Γιατί στην Κομπεχάγη αυτό που γινόταν ήταν η συνήθι απάντηση ήταν ναι, δεν γνωρίζω, θα πρέπει να διαβουλευτώ με τον Υπουργό μου και με τον Πρωθυπουργό μου. Και για να απαντήσω στον αξιότιμο κύριο Σίρβελ Περέιρα. Το ζήτημα με τα 100 δισεκατομμύρια είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για δημόσιους πόρους αυτά τα 100 δισεκατομμύρια. Είτε, είτε υπάρξουν περισσότερες δαπάνες στο, την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, είτε ε, περισσότερες δεσμεύσεις, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα από τα κρατικά ταμεία. Για εμένα λοιπόν, και το επαναλαμβάνω, απαντώντας εν μέρη και στην κυρία Χόιμπουχ, το ζήτημα δεν είναι, δεν πρέπει αυτό που θα καταλήξουμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της φτώχειας ή για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αντιθέτως, θα πρέπει συνολικά να αυξηθούν τα, ε, οι ποσά για αυτές, αυτούς τους στόχους. Ε, εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα τη σημασία ε, της αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων όπως το DCI. Αυτό το 20% για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των δωρητών. Έχουμε ορισμένες τράπεζες οι οποίες ε, έχουν δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης έχει θέσει φιλόδοξους στόχους, αλλά εμείς μέσω του blending προσπαθούμε να πετύχουμε ότι πέρα από τα δημόσια ταμεία θα υπάρξουν και ιδιωτικέ επενδύσεις. Κατά μία έννοια ιδιωτική επένδυση, οι ε, ιδιωτικές επενδύσεις βοηθούν και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ή επίσης θα πρέπει να δούμε πώς η χρηματοδότηση διαφόρων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιείται για δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Το ζήτημα του κύκλου του αζότου που αναφέρατε στη Γεωργία είναι πολύ σημαντικό. Αλλά, όπως είπατε και εσείς, ε, υπάρχουν θέματα τα οποία είναι πολύ σχετικά, πολύ συναφή με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της αποψήλωσης των δασών ή η συνδυασμός της ε, γεωργίας με τη δασοπονία. Όλα αυτά είναι μέρη μιας λύσης. Δεν γνωρίζω εγώ εάν χρειάζεται να αυξηθεί ε, η αναπτυξιακή βοήθεια. Εσείς γνωρίζετε την, αν χρειάζεται αυτή τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. βοήθειας. Έχετε δίκιο, κυρία Χουταλά, ότι το 2012 στο Φόρουμ για την Βιώσιμη Ενέργεια είχαν ε, γίνει δεσμεύσεις από τον πρόεδρο Μπαρόσο κτλ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε έναν επταετή προγραμματισμό. Και είχαμε υπολογίσει 3,6 δισεκατομμύρια, που είναι πολλά, Και αυτό ήταν η πρώτη κίνηση που ήταν απαραίτητη. Να έχουμε προγράμματα για την ενέργεια χρηματοδότηση προγραμμάτων λοιπόν σε 33 χώρε για τον εξηλεκτρισμό, για την, ε, καθαρή, για την πρόθεση της καθαρών πηγών ενέργεια, έτσι ώστε αυτό, να, να, να, υποστηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα εμείς για να ε, φτάσει, ε, να έχουν, αποκτήσουν πρόσβαση οι πιο φτωχοί άνθρωποι σε καθαρές πηγές ενέργειας. και ευελπιστώ να έρθει εκείνη η μέρα που θα ε, δοθεί, σύμφωνα με τη συμφωνία που είχαμε με τις ΗΠΑ, τα χρήματα από τις ΗΠΑ, τις οποίες θα, θα διαχειριστούμε εμείς για ε, τον εξελικτισμό ορισμένων φτώχων περιοχών. Επίσης, συμφωνώ πλήρως μαζί σας για το ζήτημα της κατανάλωσης ζωικής πρωτεΐνης. Εάν αρχίσουν και οι Κινέζοι να καταναλώνουν κρέας με τον ίδιο ρυθμό που το κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, θα χρειαζόμαστε τρεις πλανήτες για να εκτρέφουμε τα ζώα που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να πηγαίνετε εφόσον βιάσεστε κυρία Κουέν. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να είστε σύντομοι γιατί έχουμε και άλλο θέμα στη μερίσια διάταξη was already touching on, but maybe just go on, some specific. Ε, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, γιατί ζητάμε μια πενταετή αναθεώρηση και όχι μια πιο σύντομη αναθεώρηση. Νομίζω ότι ήδη εμείς ζητήσαμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψει το πακέτο αυτό ιδιαίτερα για την ενέργεια μέχρι το 2030. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε λοιπόν την προβλεψιμότητα, την απαραίτητη για αυτούς οι οποίοι πρέπει να εφαρμόσουν τις πολιτικές και εμάς και τον ιδιωτικό τομέα ε, μια περίοδος δεκαετή εν περιπτώσει και όσο σύντομη είναι η περίοδος αυτή τόσο ακριβώς, ε, τόσο ακριβώς θα μπορέσω και εγώ να δώσω μια κάποια απάντηση. Μία περίοδος λοιπόν πενταετής ή δεκαετής μπορεί να είναι ιδιαίτερος μακρά, αλλά δυόμιση χρόνια είναι πάρα πολύ σύντομο. Αλλά σε πέντε χρόνια θα ήταν ίσως ε, εύλογο να γίνει μια διάμεση αναθεώρηση. Το θετικό, κατά την απόψη μου, είναι ότι διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να ειναι ιδιαιτερως μακρα αλλα δυομιση χρονια ειναι παρα πολυ συντομο αλλα σε πεντε χρονια θα ηταν ισως ευλογο να γινει μια διαμεση αναθεωρηση το θετικο κατα την αποψη μου ειναι οτι διαπιστωνουμε οτι τα κρατη μελη της ευρωπαικης ενωσης θελουν να αυξησουν τη χρηματοδότηση από του κρατικού προπολογισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγή και για την βοήθεια των πλέον ευάλωτων ομάδων, των πλέον φτωχών. Αυτό θα γίνεται με τη μορφή κατά κύριο λόγο επιδοτήσεων προ τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρες, αλλά επίσης πρέπει να βρούμε μια ισορροπία έτσι ώστε τα χρήματα να κατευθυνθούν ε, χρηματοδοτικά μέσα που μας επιτρέπουν να υπάρξει και εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αποστείλουμε τα χρήματα και σε περισσότερες χώρες. Επίσης, συμφωνώ ότι χρειάζεται να ε, ενισχυθεί η λογοδοσία όταν υπάρχει συμμετοχή ε, του ιδιωτικού τομέα, ιδίως χρηματοδοτικά μέσα τύπου blending. Είναι πολύ διαφορετικό βέβαια το ζήτημα της άμεσης χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, και η λογοδοσία είναι πολύ πιο δύσκολη. Έχει αναφερθεί η δυνατότητα των λεγόμενων πράσινων επιδοτήσεων, green bonds, ή και άλλα χρηματοδοτικά καινοτόμα μέσα, τα οποία βέβαια πρέπει να τα εξετάσουμε ε, λαμβάνουμε τις σχετικές εισηγήσεις από τους ειδικού, έτσι ώστε να έχουμε και μια εξασφάλιση ότι τα, έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο είναι πράγματι φιλικά προς το περιβάλλον. Οκ. Η επόμενη ομιλήτρια παρακαλώ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να, να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Κυρίως κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο πρέσβης Ροντόλφη, αν και έφυγε δυστυχώ, θα ήθελα να πω ποια είναι η άποψη των μη κυβερνητικών οργανώσεων όσον αφορά τα 100 δισεκατομμύρια ε, μέχρι το 2020 και αν αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια χρήματα ή όχι. Αντιλαμβανόμαστε και και καταλαβαίνουμε ότι στην συμφωνία της Κοπενχάγης είχε καταγραφεί ότι αυτά τα 100 δεν θα είναι μονοκρατικά, ωστόσο η θέση των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ότι θα πρέπει να είναι κρατικά, γιατί είναι άγνωστη πόσο μεγάλη, θα είναι, πόσο μεγάλη μικρή θα είναι η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα. Και είναι κρίσιμη σημασία να βρεθούν τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Τώρα, εάν αυτά θα είναι χρήματα πρόσθετα προς την ODA, την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό δεν έχει συμβεί, αλλά η θέση μας είναι ότι αφού η κλιματική αλλαγή είναι μια επιπλέον, μια ξεχωριστή ε, πρόκληση, θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστή και επιπλέον χρηματοδότηση. Αφού αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι εξαιρετικά μη φιλόδοξοι. Δηλαδή στην Αντισάμπαμπα είδαμε ότι τα πράγματα δεν προχώρησαν όσο θα θέλαμε. Συμπερασματικά το ζήτημα είναι πώς θα αυξηθεί συνολικά η χρηματοδότηση. Και πιστεύουμε ότι στο μέλλον οποιοδήποτε έργο χρηματοδοτείται μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να εξετάζεται αν είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αν συνεισφέρει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είτε αυτό γίνεται μέσω της ODA, είτε μέσω ε, επενδυτικών τραπεζών, αλλά συνεχίζει να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, η οποία κατευθύνεται προς έργα μη φιλικά προς το περιβάλλον ακόμα και σε έργα, για παράδειγμα, για χρήση άνθρακα. Επομένως, από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι αφενός πρέπει να στηθεί η κρατική χρηματοδότηση, αλλά και αφετέρου θα πρέπει να υπάρξει ε, ευαισθητοποίηση στο εθνικό και στο τοπικό επίπεδο για τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ε, των έργων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Όταν λέγεται ότι οι προπολογισμοί δεν επαρκούν, αναρωτιέται κανείς και τότε πώς καταφέρνουμε να υποδοτούμε τα ορυκτά καύσιμα. Όταν κοιτάμε τα δισεκατομμύρια που ε, δίνονται για επιδοτήσει ορεικτών καυσίμων, ε, είναι λογικό να ασκεί κανεί κριτική για να αναρωτιέται. Και πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο κάθε κράτου μέλου. Κάθε κράτο μέλο πρέπει να σκεφτεί τελικά τα χρήματα που δίνει πηγαίνουν προ έργα τα οποία συνεισφέρουν στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Τετιάνα, έχετε πολύ λίγο χρόνο στη διαθέσή σα. Θα είμαι σύντομη γιατί περισσότερα ζητήματα έχουν ήδη απαντηθεί. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ξεχωρίσουμε την ανάπτυξη από τη μία και τις κλιματολογικές αλλαγές από την άλλη. Απλά οι κλιματολογικές αλλαγές επιβαρύνουν τις προκλήσεις των τρίτων χωρών. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι ευαίσθητη στο κλίμα και το κομμάτι το οποίο ας έχει σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές θα επιβαρυνθεί στο μέλλον. Λυπάμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, λέει η Πρόεδρος. Και τελευταίο θέμα είναι το λεγόμενο question time. Το 24 μιλήσαμε για τις κλιματολογικές αλλαγές και για τη διάσκεψη για τη μείωση των ε, συνεπειών και των ζημιών ε, από, τα φαινόμενα των κλιματολογικών αλλαγών. Ο κύριος Γκουέρο Σαλόμ είχε θέσει ένα ερώτημα στην Επιτροπή. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ντολανουά από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, πάνω από 10 λεπτά δεν έχουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Γκοέρο Σαλόμ για το θέμα της δράσης της Σανγκάη, για το διεθνές πλαίσιο, δηλαδή για τη μείωση των κινδύνων που υιοθετήθηκε στην Ιαπωνία. Τον προηγούμενο Μάρτιο παίξαμε ένα σημαντικό ρόλο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις της Σανγκάη και για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Όπως είπατε στην ερώτησή σας κύριε Γκουερέρο Στολόμ, έχει σημασία να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα ανάμεσα στις αποφάσεις της Σανγκάη, στις αποφάσεις για την ατζέντα του 2030 και στις διαπραγματεύσεις για τις κλιματολογικές αλλαγές. Το πρόγραμμα δράσης της Σανγκάη αναγνωρίζει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη διαχείριση των κινδύνων των καταστροφών, στην αηφορία και στην ατζέντα η οποία περιλαμβάνει πολλούς δείκτες όπως η ανθεκτικότητα, η μείωση των κινδύνων, οι ανθεκτικές υποδομές, η προστασία της υγείας και της εκπαίδευσης. Πρέπει λοιπόν οι δείκτες αυτοί να συνδέονται με τους δείκτες που αναπτύσσονται για το πλαίσιο της δράσης της Σανγκάη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτούς τους στενούς δεσμούς. Μία από τις προτεραιότητες της Σανγκάη είναι η μείωση των κινδύνων στα πλαίσια των πολυμερών και διμερών προγραμμάτων για την ανάπτυξη. Είναι μία από τις προτεραιότητες και του πλαισίου της Άντης και προσπαθούμε εμείς να συνδέσουμε τις δύο διαδικασίες. Και τέλος, Υπάρχει ένα στενός δεσμός ανάμεσα στη διαχείριση των κινδύνων από τη μία και τις κλιματολογικές αλλαγές από την άλλη. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την συνοχή ανάμεσα στην προσαρμογή για τις κλιματολογικές αλλαγές και τη διαχείριση των κινδύνων. Εθνική στρατηγική για τις κλιματολογικές προσαρμογές, ο ρόλος των ασφαλιών και ο ρόλος τον οποίο πρέπει να έχει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Αυτή είναι προτεραιότητα της COP21. Πώς να καταλήξουμε δηλαδή σε συγκεκριμένες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε και τις κλιματολογικές αλλαγές και την μείωση των κινδύνων. Συνεργαζόμεθα με την Γαλλική Προεδρία και με την Περουβιανή επίσης σε σχέση με την Λατινική Αμερική για τις μελλοντικές δράσεις τις οποίες προβλέπεται να αναπτύξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα δημοσιεύσει ένα πρόγραμμα δράσης στα πλαίσια του 2016, μέσα στο 2016. Προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι υπάρχουσες πολιτικές που συμμετέχουν στη μείωση των κινδύνων. Ε, πολιτική προστασία, αύξηση της ανθεκτικότητας των υποδομών, και σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε επίσης και τον τρόπο με τον οποίο η περιβαλλοντική πολιτική, η πολιτική στην υγεία, η πολιτική στην πολιτιστική κληρονομιά και την εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει. Έχουμε ανακοινώσει επίσης ότι θα θέσουμε σε λειτουργία και την Ατζέντα 2030 για την αηφόρο ανάπτυξη. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει μια πρωτοβουλία η οποία ε, θα λάβει υπόψη τους στόχους ε, της ε, αηφορίας των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσουμε επίσης και με την εφαρμογή του προγράμματος δράσης ανθεκτικότητας που περιλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες που θα αποκαταστήσουν στενούς θεσμούς ανάμεσα στη μείωση των κινδύνων και στην προσαρμογή στις κλιματολογικές αλλαγές. Διάφορες πρωτοβουλίες όπως JCCR, SHARE ε, και Azure. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Στα πλαίσια αυτών των νέων πρωτοβουλειών που αναπτύξαμε ήδη ε, και θα συνεχίσουμε πριν το 16. Ο Γκουερέρος Σαλόμ σύντομα. Λοιπόν, ευχαριστώ για μια πλήρη θα έλεγα και ευρύτατη απάντηση από πλευράς ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ήθελα να ακριβώς να μάθω τι ακριβώς βάζει σε επαφή, θέτει σε επαφή τη Σανγκάη με την Άντις και με τη Νέα Υόρκη και τώρα με το Παρίσι για τις κλιματολογικές αλλαγές. Εποφελούμε λοιπόν από την ευκαιρία για να πω ότι υιοθέτησε η Επιτροπή την έκθεση του Κοινοβουλίου για την ανθρωπιστική συνάντηση κορυφής στην Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στην πρόταση της για τη μείωση των κινδύνων και να τη συνδέσει με την συνάντηση κορυφής και την συζήτηση για τις προληπτικές δράσεις που μπορεί να επηρεάσουν και τις ανθρωπιστικές κρίσεις όσαν οφείλονται βέβαια σε φυσικές καταστροφές. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Αυτά ε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί. Στα διάφορα ε, δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι να σας ευχαριστήσω ότι στην Ολομέλεια θα γίνει συζήτηση για τη βοήθεια στην Αφρική και για την συνάντηση κορυφή στη Βαλέτα. Η επόμενη συνάντησή μας είναι την 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ την διευμηνία. Χρησιμοποίησαμε λίγα λεπτά από τα διαθέσιμα.